Uh, dear colleagues, we're going to make a start. We've paused. Ξεκινήσουμε συνάδελφοι. Περιμέναμε μπας και έρθουν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη σήμερα και εν ώψη της ε, συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών σήμερα και της ε, ημερήσιας διάταξη που έχουμε για τα θέματα μετανάστευσης. Έχουμε πολλά σημεία στη μέση διάταξη. Προσοχή. Θα ακούσουμε την Επιτροπή για μια παρουσίαση για το δεύτερο μεταναστευτικό πακέτο που παρουσίασε σε 9 Σεπτεμβρίου και Πρόεδρος Γιώργη. για ό,τι αφορά τα προσωρινά με την προστασία διεθνού, για την, στο δομέα της διεθνούς προστασίας για Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία, σημείο 5 που ψηφίσαμε στην Ομιλία την, πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη, η Προεδρία είναι έτοιμη να ενημερώσει την Επιτροπή μας για την κατάσταση των συζητήσεων στο Συμβούλιο τις τελευταίες μέρες εν ώψη και της, ε, του Συμβούλου Υπουργών Εσωτερικών απόψη. Η Προεδρία ζήτησε να γίνει και κλεισμένο το, το θέμα αυτό γιατί οι συζητήσεις προχωρούν ακόμα. Ε, την, όπως ξέρετε την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια άτυπη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για τα θέματα της ε, μετεγκατάστασης. Οι περισσότερες ε, ομάδες υποστήριξαν να γίνει και κλεισμένο το θεών αυτή η ενημέρωση και θα γίνει στις 11.30. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Ένα διαδικαστικό κύριε Βαμπέρ. Μία ερώτηση για το σημείο 5, Πρόεδρε. Γιατί γίνεται η ενημέρωση και κρισμένο των θυρών, γιατί δεν μπορεί να ακούσει το κοινό τη σχετική συζήτηση. Εγώ είμαι αντίθετο. Εγώ είμαι αντίθετη με αυτό το θέμα. Για το ίδιο θέμα και εσείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ενίσταμαι στην ε, συζήτηση του σημείου αυτού και κλεισμένων των θυρών. Την περασμένη εβδομάδα σε μια έκτακτη συνάντηση υποστηρίξαμε στο Κοινοβούλιο την πρόταση της Επιτροπής. Δεν θεωρώ ότι αυτό συνάδει με μια συζήτηση και κλεισμένων των θυρών. Οι πρόσφυγες και οι άσυλο στο ένα μεταξύ ε, βρίσκονται παντού στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει με ανοιχτέ διαδικασίες. Να απαντήσω και στις δύο, λέει ο Πρόεδρος. Πρόκειται για ενημέρωση όχι συζήτηση και κλεισμένων των θυρών για μια σειρά ζητημάτων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Η πλειοψηφία των συντονιστών συζήτησαν και δέχτηκαν να υπάρξει ενημέρωση και κλεισμένων των θυρών. Δεν γίνεται ενημέρωση ε, θεμάτων που συζητούνται ακόμα. Εγώ προτείνω να συνεχίσουμε ε, και κλεισμένων των θυρών. Τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά βεβαίως, αλλά πρόκειται για ενημέρωση, όχι για συζήτηση. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ε, ενστάσεις ή διαδικαστικά, να προχωρήσουμε. Σημείο 2. Δυστυχώς, συνάδελφοι, δεν υπάρχει διερμηνία στα κροατικά, δανέζικα, Ιρλανδικά και Λετωνικά. Θα έχουμε Κροατικά και Ιρλανδικά, δεν θα έχουμε ούτε και αύριο. Τώρα, ως εισηγητές. Ο κύριος Κίρκοπ, εισηγητής για την έκθεση μόνιμη κρίση, ένας μηχανισμός μόνιμης ε, κατάσταση βάση του Δουβλίνου θα ήθελα να ζητήσω να υποστηρίξετε την σύσταση της των ιστών, ούτω και γένετο. Σημείο 3. Στις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Θα υπάρξει ηλεκτρονική ψηφοφορία σήμερα στις 5 ε, το απόγευμα, να έχετε μαζί σας τις κάρτες σας. Προχωρούμε. Κοινή συζήτηση. Όπως σας είπα, Ξεκινούμε με το σημείο 3. Ο μηχανισμός κατάσταση λόγω κρίσεως και μηχανισμοί για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτηση διεθνούς προστασία που υποβάλλεται από κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος από υπήκο τρίτης χώρας ή ηθαγενή. Κάποιες πληροφορίες μόνο για το πώς θα γίνει η συζήτηση θα υπάρξει μια παρουσίαση από την Επιτροπή για το δεύτερο μεταναστευτικό πακέτο όπως ανακοινωθήκε στις 9 Σεπτεμβρίου από τον πρόεδρο Γιούνκερ. Θα δώσω κατόπιν το λόγο στην Επιτροπή, κατόπιν στα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να μιλήσουν, ξεκινώντας από συντονιστές και σκιώδεις εισηγητές για την ολιστική προσέγγιση μετανάστευση. Κατόπιν θα ξεκινήσουμε με δύο παρατηρήσει, με δύο παρουσιάσεις για δύο νομοθετικά κείμενα. Ζητώ λοιπόν καταρχάς από την Επιτροπή να μα παρουσιάσει το σχέδιο κανονισμού για τον μόνιμο μηχανισμό με την κατάσταση λόγω κρίσεως και το σχέδιο κανονισμού για το σημείο 4 της ασφαλής χώρας καταγωγής. Κατόπιν θα μιλήσουν οι συνάδελφοι, οι συντονιστές και, τα, και οι συνάδελφοι. Σας έχω μπερδέψει λίγο συνάδελφοι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ξεκινούμε λοιπόν παρουσιάσεις από την Επιτροπή. Ο κύριος Ρίσε, παρακαλώ. Κατόπιν το λόγο θα λάβουν οι συντονιστές και τα μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, θα ξεκινήσετε πρώτα με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και μετά με το κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής και μετά τη συζήτηση θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα θέματα. Κοιτάξτε, αν μείνετε για τη συζήτηση, το δεύτερο μέρος της κοινή συζήτησης, θα ζητήσω να γίνει αυτή η παρουσίαση και μετά το τρίτο μέρος θα μιλήσουμε για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της περιοχής. Και θα μιλήσουμε λοιπόν, ε, θα χωριστεί συζήτηση σε τρία μέρα. Παρακαλώ λοιπόν. Για μιλήσετε, ε, θα μιλήσετε καταρχά για τον <clears throat> μηχανισμό κατάσταση. Όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, προτείναμε ένα μόνιμο πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό το Σεπτέμβριο. Προτείναμε μια ε, κάναμε μια πρόταση να μετεγκατασταθούν ε, 120.000 άτομα. Ο στόχος είναι να αποφύγουμε τα όσα βιώσαμε φέτος το καλοκαίρι και να καταβάλουμε μία προσπάθεια να βρούμε μία κατάλληλη λύση με ένα πρόβλημα προς, ε, μόνιμης μετεγκατάστασης. Τη στιγμή που υπήρξαν δύσκολες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο θα θέλαμε να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης, ένα πρόγραμμα που θα αναπτύσσεται κάθε φορά που υπάρχει μία κρίση. Κάθε φορά θα βρίσκεται μία λύση με ένα διαφορετικό τρόπο κατανομής, με διαφορετικό διαφορετικό τρόπο διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών μελών. Προτείνουμε το άρθρο 78 παράγραφος 2 της συνθήκης επιμένω γιατί όπως γνωρίζετε το άλλο πρόγραμμα δίνει ε, εξουσία, πλήρη εξουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά επανερχόμεθα στη συναπόφαση. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο να στραφούμε προς αυτό το πλαίσιο, προς αυτό το πρόγραμμα. Προτείνουμε την ε, κατεξουσιδότηση πράξης για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμός μεταγκατάστασης όταν ε, θεωρούμε ότι η κατάσταση μπορεί να αποβεί κρίσιμη για μία χώρα μέλος. Όταν δηλαδή ασκούνται ακραίες πιέσεις σε μία χώρα μέλος, ακόμα και σε περιπτώσεις που το σύστημα χορήγησης ασύλου λειτουργεί σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες. Το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά με χώρες μέλη που πληρούν τις προποθέσεις ή κάνουν το καθήκον τους, είναι για περιπτώσεις που ασκούνται πιέσεις ακόμα και όταν μία χώρα μέλος κάνει αυτά που καλείται να κάνει. Δημιουργήσαμε ένα μηχανισμό κατανομής που είναι παρεμφερής με αυτόν που προτείνουμε το, στα προσωρινά προγράμματα κατάσταση και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί σήμερα το ε, απόγευμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις περιπτώσεις που μια χώρα μέλος αρνείται αυτό το ε, πρόγραμμα. Έχουμε θέσει τέσσερα κριτήρια πληθυσμός, το ΑΕΠ, ε, το 40% στο πρώτο, 40% στο δεύτερο, αριθμός τούντων άσυλο κατά κεφαλή 10%, και ανεργία 10%. Και υπάρχει ένας μηχανισμός σύζευξης για να αποφύγουμε τα ποσοστά αυτά είναι, να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την κατανομή τους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια εξισορροπημένη πρόταση και εμείς θα λέγαμε να την εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατόν ασκούνται πάρα πολλές αντιστάσεις σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Δεύτερη νομοθετική πρόταση. Η δεύτερη αφορά τις ασφαλείς χώρες καταγωγής ή ε, όπως γνωρίζετε οι χώρες μέλη μπορούν σύμφωνα με το περί ασύλου και κτημένο να έχουν τους δικούς τους εθνικούς καταλόγους. 12 ε, χώρες έχουν ε, καταλόγους με ασφαλείς ε, χώρες καταγωγής. Υπάρχουν βέβαια διαφορές και θεωρούμε ότι η ροή των τούντων άσυλο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μία επιτάχυση των διαδικασιών σε ό,τι αφορούν τα άτομα που προέρχονται από τη Δυτική Όχθη εκεί το ποσοστό είναι χαμηλό. Θα ήθελα να επιμείνω ότι όταν προέρχεται κανείς από μια χώρα που βρίσκεται στον κατάλογο ασφαλών χωρών, δεν σημαίνει ότι δεν θα τύχει επεξεργασία ή αίτηση ασύλου. Όλοι θα αξιολογηθούν ανάλογα ε, με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά αν κάποιος, ε, κάποιου χώρα ανήκει στις ασφαλείς χώρες καταγωγής, η διαδικασία θα επιταχυνθεί. Έχουμε προτείνει 7 χώρες να συμπεριληφθούν σε αυτό τον κατάλογο. Ε, ε, ε, Φύρο, σε Σερβία, Τουρκία, Αλβανία. Συνεπώς θεωρούμε ότι πέντε υποψήφιες χώρες θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρωπινά δικαιώματα, σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων. Και εδώ προστίθεται η ε, Ζεγοβίνη και το Κόσοπο. Και αυτό με βάση το γεγονός ότι έχουν ένα χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για θέματα ασύλου. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι 7 αυτέ χώρε πληρούν τι προποθέσει ε, που έχουν τεθεί από την οδηγία για το άσυλο και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασφαλεί χώρε καταγωγή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ελέγχει εκ του σύνεγγυ την κατάσταση σε αυτέ τι χώρε. Αυτό που προτείναμε είναι έναν ρυθμό, ένα ε, ε, γρήγορο μηχανισμό για να βγει, για να απομακρυνθεί μια χώρα από τον κατάλογο. Εμείς λέμε να υιοθετήσουμε τον κατάλογο με συναπόφαση, αλλά να, για να αφαιρεθεί μια χώρα από τον κατάλογο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ας πούμε, αν ένας επικεφαλής κράτους ε, υιοθετεί χτίσει μία απόφαση που να στρέφεται κατά της ελευθερίας του τύπου ή των μειονοτήτων. Αυτό θα πρέπει αυτόματα να μας οδηγήσει στη διαγραφή της χώρας από την ασφαλή χώρα ε, καταγωγής. Έχουμε και ένα μηχανισμό ανάκλησης. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί πάντοτε να διτεθεί σε μια τέτοια ανάκληση. Αυτό δεν γίνεται στα πλαίσια της συναπόφασης για να διαγραφεί η χώρα, γίνεται μια ανάκληση της κατεξουσιοδότηση πράξης. Και αν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η ανάκληση θα πρέπει να είναι μόνιμη, τότε περνάμε στην νομοθετική διαδικασία μέσω της τακτικής διαδικασίας. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κατάλογος για να ανακληθεί προσωρινά μία χώρα από τον κατάλογο. Το γεγονός ότι μια χώρα είναι, θεωρείται Ασφαλή χώρα καταγωγή, ε, δεν συνεπάγεται ότι δεν ατύχει επεξεργασία το αίτημα χορήγηση ασύλου. Ε, οι αιτούντε από τη Δυτική Όχθη είναι το 17% των αιτήσεων. Συνεπώ αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα το σύστημα ασύλου και θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα άτομα που σαφώς χρειάζονται διεθνή προστασία και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις που γίνονται σε ό,τι αφορά την, τις αιτήσει που υποβάλλονται για χορήγηση ασύλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε κατευθείαν στους συντονιστές να τοποθετηθούν αυτοί σχετικά με αυτό το μηχανισμό μετεγκατάστασης. Παρακαλώ, η Birgit. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την άποψη ότι πρέπει να δώσουμε μια διάρθρωση σε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους. Εφόσον μιλάμε για το μηχανισμό κατάσταση πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση μοιάζει να είναι χαοτική όσον αφορά τις ροές μεταναστών. Και είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ένα τμήμα αυτού του μηχανισμού κατάστασης ε, δεν αφορά μόνο το ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αλλά και το ότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε όλοι οι μετανάστες όπου κι αν φτάνουν τα καταγράφονται. Να υπάρχουν τα σημεία καταγραφής έτσι ώστε όπως σας είπα να καταγράφονται όλοι οι μετανάστες και μετά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πολύ καλή βάση μετεγκατάστασης. Πάμε τώρα στον κατάλογο των, ε, με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα ότι αν ξαφνικά τα μέσα ασκήσουν πίεση, η χώρα αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Παράλληλα διαβάζω, υπάρχουν κάποιες χώρες ε, στους ε, καταλόγους ε, και οι δημοσιογράφοι ήδη ασκούν πίεση και ρωτώ γιατί εξακολουθούν να βρίσκονται στον κατάλογο και να προσθέσω κάτι άλλο. Ωραίο είναι να λέει κανείς ότι κάποιες χώρες είναι υποψήφιες χώρες και οφείλουν να καλύπτουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Όμως δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό διότι στην πραγματικότητα δεν καλύπτουν τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης. Άρα δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί το να λέμε ότι στα χαρτιά ε, καλύπτουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης αυτό μπορεί να οδηγήσει και στο συμπέρασμα από δική σου πλευράς γιατί δεν μπαίνουμε κι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν. Και μία τελευταία παρατήρηση. Όταν μιλάμε για ταχύτερες ε, διαδικασίες. Αυτό σχετίζεται με τις οδηγίες που περιλαμβάνει το πακέτο περιασύλου σχετικά με την υποδοχή ε, και τις άλλες διαδικασίες. Αν λοιπόν θέλουμε επιτάχυνση των διαδικασιών, το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει ε, την ε, οδηγία περί χορήγησης ασύλου. Δηλαδή να εξετάζουν το αίτημα ασύλου. Αν όχι, τότε πώς είναι δυνατόν να συζητάμε διαδικασία επιτάχυνσης ε, αν δεν υπάρχει σαφή διαδικασία. Κατόπιν τούτου, μερικές φορές πρέπει να εξετάζουμε και να διασφαλίζουμε όχι ένα μέτρο, αλλά το σύνολο των μέτρων να εξασφαλίζουμε ότι όλα τα μέτρα εφαρμόζονται σωστά έτσι ώστε στη τελική ανάλυση να καταλήγουμε σε ένα καλό πακέτο και όχι οι ψηφίδες ενός μουσιακού οι οποίες ε, δεν παίρνουν τίποτα. Πρόεδρος, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις, ε, η Κορνίλια τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να ε, ληφθούν μέτρα εκ μέρους της ε, Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι πολύ καλό που μας συμπεριλαμβάνουν και εμάς στη συζήτηση. Θα ήταν απαράδεκτο να μην γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά το μηχανισμό μετεγκατάστασης, πράγματι είναι αλήθεια ότι σε αυτόν πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερες χώρες. Εγώ αυτό το βρίσκω σωστό και επίση το βρίσκω σωστό να υπάρχει και μία κλίδα κατανομής. Αλλά μία κλίδα κατανομής η οποία ε, αφορά κριτήρια τα οποία όμως ορίζουν τα κράτη-μέλη, αυτό δεν το βρίσκω και πολύ λογικό, γιατί δεν έχει νόημα να μοιράσει κανείς ε, δια του 28 αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία, όσον συζητάμε, στην ύπαρξη των μεγάλων κοινοτήτων, με λίγα λόγια δηλαδή. Στη Γερμανία, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη συριακή κοινότητα, άρα θα είχε νόημα σε αυτή την ε, περιοχή να εγκατασταθούν κάποιοι άνθρωποι. Αλλού όταν δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κοινότητα δεν έχει νόημα να πάνε εκεί οι πρόσφυγες. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και να δούμε και λιγάκι ακριβώς το θέμα των ε, προσφύγων. Διότι μην ξεχνάτε στην Ευρώπη θα συνεχίσουν οι μετακινήσεις. Αυτή είναι η πρώτη κριτική που ασκώ. Και το δεύτερο είναι το Ό,τι και αν γίνει πρέπει να είναι δεσμευτικό. Γιατί αν ε, όλα είναι δεσμευτικά, τότε αυτό το προαιρετικό μηχανισμό τον βρίσκω ανεύθυνο. Κάτι άλλο, αυτό που επίσης πρέπει να ζητήσουμε είναι ένα κοινό σύστημα ασύλου για την εναρμόνιση. Η εναρμόνιση του ε, συστήματος ασύλου, γιατί μερικά κράτη δεν έχουν καθόλου σύστημα, αυτό είναι απαράδεκτο. Και νομίζω αυτό δεν φαίνεται αρκετά την ε, πρόταση που έχει υποβληθεί. Και κάτι άλλο επιτρέψτε μου να πω. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι απόδειξη του ότι έχει πεθάνει το Δουβλίνο. Το σύστημα του Δουβλίνου έχει πεθάνει. Μπορούμε βέβαια να το αναστήσουμε, μπορούμε να γράψουμε ότι ε, στο πλαίσιο, ότι διαπραγματευόμεθα στο πλαίσιο του Δουβλίνου, αλλά αυτό σας λέω έχει πεθάνει και αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ό,τι και να κάνουμε, το κατά πόσον τα ακολουθήσουμε το βιβλίο ή όχι, υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Και κάτι άλλο. Γνωρίζω αρκετά καλά τα Δυτικά Βαλκάνια, αρκετές χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Και πρέπει να σας πω ότι δεν ε, πιστεύουν ότι πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Μερικά αγωνίζονται να επιβιώσουν, όπω το Κοσμοπέδιο και θα με ενδιαφέρει να ακούσω από την Επιτροπή με βάση ποια κριτήρια προχωρήσατε για να ορίσετε ότι αυτά τα κράτη είναι πράγματι ασφαλή για αυτές τις χώρες. Ποια είναι τα κριτήρια και τι κάνετε σε σχέση με τους Ρωμά. Για εξηγήστε μου, το Κωσυφοπέδιο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν πια διώξεις εναντίον των Ρωμά, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση εναντί τους. Και αν μπορείτε να μου πείτε τη λύση θα σας προτείνω στη Γερμανία για βραβείο ειρήνης. Ίσως ε, να υπάρχει κάποιος ε, μηχανισμός ε, αναστολής. Εγώ θα ήθελα να τον ετηθώ αυτό κυρίως για τους Ρωμά του Κωσυφοπεδίου. Με όλα αυτά που λέμε, τελικά το δικαίωμα για άσυλο και για αξιοπρεπή ζωή, νομίζω το δικαίωμα αυτό υπονομεύεται και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να το επιδιώξουμε. Σας ευχαριστώ. Σεσίλια Βίξτο, επόμενη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξεκινώ πρώτα με την έννοια του καταλόγου των ασφαλών χωρών. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Επιτροπή που υπογραμμίζει πάντα ότι κάθε εφαρμογή της διάταξης αυτή πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό του ατομικού δικαιώματος στο άσυλο και ότι ο κατάλογος, η έννοια του καταλόγου των ασφαλών χωρών καταγωγής δεν περιορίζει το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα. Χαίρομαι που το, το, το τονίζει πάντα η Επιτροπή και θα ήθελα να το ξανακούσω ως εισηγήτρια για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου την περασμένη θητεία δουλέψαμε πολύ σκληρά και πρέπει να σας πω ότι εγώ πάνω απ' όλους είμαι ευτυχέστερη που βλέπω ότι ο κανονισμός Δουβλίνου δεν μας βοηθά στην κατάσταση αυτή. Αντιμετωπίζουμε κάποιες από τις προφανείς πλέον αυτού του νομικού κειμένου. Είναι θλιβερό απλώς το ότι διαπιστώνουμε μόνο τώρα ότι χρειάστηκε δηλαδή αυτή η τεράστια κρίση για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να καταλάβουν τα λάθη τους. Και ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη ζουν σε μια μορφή άρνησης ακόμα. Πρέπει να ξυπνήσουν και να δουν την πραγματικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να τους περάσω. Τρεις ερωτήσεις έχω σήμερα προς την Επιτροπή για να διευκρινίσω μια σειρά προτάσεων, για να καταλάβω, καταλάβω, καταλάβω καλύτερα. 33α πρώτα πρώτα. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 6 αναφέρει μια διάταξη που λέει ότι ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να μετεγκατασταθεί βάσει του, κανον, του επίγοντος κανονισμού θα ξεπεράσει το 40% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο κράτος μέλος αυτό κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν την έγκριση της κατεξοδότησης πράξεως. Αν καταλαβαίνω καλά τη διαδικασία, αυτό μπορεί να κρατήσει μια διετή περίοδο. Ας δεχθούμε μια υποθεωτική μαθηματική περίπτωση. Δεν θέλω να σας κουράσω, απλά ε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει τον κίνδυνο να κάνει τη μετεγκατάσταση κάπως αδύναμη για να βοηθήσει πραγματικά ένα κράτος που χρειάζεται βοήθεια. Αν δείτε τους παράγοντες αυτούς, συνδυάζοντας με την πρόταση αυτή, θα καταλάβετε ότι σε κάποια περίπτωση μπορεί να μετακατασταθούν πολύ λίγοι εν τέλει. Επίσης, ποιος είναι ο ρόλος του ΕΑΖΟ στην επιλογή των ατόμων που θα μπουν σε διαδικασία μετακατάστασης. Αν κατάλαβα την πρόταση της Επιτροπής, η ΕΑΖΟ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο. Κατά την άποψή μου, προσπαθήσαμε να το δούμε αυτό σε μακρό χρονικό διάστημα και προτείνουμε στην ομάδα μου έναν ισχυρότερο ρόλο για την ΕΑΖΟ. Ίσως και την ανάθεση σε αυτήν της ευθύνη να κάνει την διαδικασία επιλογής στην συνεργασία με τις εθνικές αρχές γιατί αυτό θα επιτρέψει σε κράτη-μέλη που δέχονται ε, μετεγκαταστημένους ετούντες άσυλου να είναι βέβαιοι ότι δεν έγινε επιλογή από τρίτους. Μια τελευταία παρατηρήση θα ήταν σκόπιμο να μας φωτίσει Επιτροπή για την πιθανή συμμετοχή συνδεδεμένων κρατών με το Δουβλίνο, Δανία, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία. Θα επιλέξουν ή όχι να εφαρμόσουν τον κανονισμό του Δουβλίνου μετά την αλλαγή. Αν υιοθετηθεί ο μηχανισμός μετακατάστασης λόγω κρίσεως σημαίνει ότι οι χώρες αυτές θα λάβουν και αυτές ετούντες βάσει του κανονισμού. Θα πρέπει να πληρώσουν το 0,002% της συμφοράς τους στο ΑΕΠ σε περίπτωση που δεν δεχθούν να μετάσχουν στο σύστημα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ε, ακούμε τις απόψεις επιτοπής μετά από κάθε μία από τις τρεις ε, συζητήσεις. Τα υπόλοιπα μέλη. Η Σοράγια. Ευχαριστώ. Βλέποντας την κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα είναι σαφές ότι το Δουβλίνο πάει πια. Και εδώ είναι η Επιτροπή να το καταλάβει και να το αναθεωρήσει. Ελπίζω να γίνει κατανοητή, κατανοητό ότι η μόνη λογική λύση είναι η κατάργηση του Δουβλίνου και η δυνατότητα στον κόσμο, να, στους ετούντες, να επιλέξουν που θα ζητήσουν προστασία. Ο μηχανισμός ε, με την κατάσταση είναι βέβαια ουσιαστικός διότι υπάρχουν άτομα που ξεκινούν σε κάποια κράτη-μέλη και φωτώνουν τη διαδικασία σε αυτά. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη πρέπει να δεχθούν την ευθύνη τους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι λογικό να εξαγοράσεις την ευθύνη αυτή πληρώνοντας χρήματα. Μία ερώτηση λοιπόν που μπορώ να θέσω είναι ποιοι λόγοι είναι αυτοί που δικαιολογούν την αίτηση ενός κράτους να εξαιρεθεί. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχω απλά χρήματα. Μια σοβαρή έλλειψη στην πρόταση είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα του ατόμου. Ο κάθε ετών, ο κάθε πρόσφυγας δεν φαίνεται να έχει δικαιώματα. Ένας ετών που δεν έχει δικαιώματα μπορεί να απελαθεί ακόμα και αν υπάρχει καλύτερη πρόθεση. Άλλη παρατήρηση λοιπόν, πώς θα λάβει υπόψη η πρόταση αυτή τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων που πηγαίνουν προς μετεγκατάσταση για να μην υπάρξει παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Για τις ασφαλείς χώρες καταγωγής, σε συνέχεια αυτό που είπε η Κορνέλια, οι χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, κατά την άποψή μου, σε τρεις ή σε τέσσερις από αυτές τις επτά χώρες που αναφέρονται η ασφάλεια δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά τους Ρωμά. Βεβαίως οι Ρωμά δεν πυροβολούνται, δεν βομβαρδίζονται, βοβαρδιζονται αλλα ζουν σε συνθήκες που δεν αρμόζουν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτές είναι χώρες στις οποίες κατοικούν ε, κατοικούσαν, ε, υπάρχουν χώρες που κατοικούσαν για γενιές, αλλά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους έχουν αναγκαστεί να φύγουν. Ε, πώς εξασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου τους γίνεται με δίκαιο και σωστό τρόπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κλείσω τον κατάλογο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Έχω τον κατάλογο με που θέλουν να μιλήσουν. μάλλον ε, μιλιών. Ε, Ευχαριστώ. Πολλά από όσα σκόπευα να πω ήδη υπόθηκαν, δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω και πάλι. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω ότι σε ό,τι αφορά το μηχανισμό μετεγκατάστασης Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι προτιμήσεις, οι επιθυμίες των μεταναστών. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν συνυπολογίζεται. Μιλάμε για επανένωση των οικογενειών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι επιθυμίες του μετανάστη. Αν ε, Βεβαίω δεν αμφισβητείται η σύμβαση του Δουβλίνου, αυτό σημαίνει ότι απέχουμε πολύ από μία λύση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Θα πρέπει σταδιακά να καταργηθεί η σύμβαση του Δουβλίνου, θα πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο θέμα. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον κατάλογο αυτό. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην κατάσταση το Ρωμά στις χώρες αυτές. Αν κοιτάξουμε επίσης τις προπαρασκευαστικές εργασίες ε, ε, που έγιναν, θα δούμε ότι το Συμβούλιο δεν θεωρούσε ότι η Τουρκία θα έπρεπε να παραμείνει σε αυτό το κατάλογο. Το 23,1% των αιτήσεων ασύλου πρόκειται από άτομα που διέσχισαν την Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν. Η Τουρκία δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Ευχαριστώ. Ε, εγώ θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι σε ό,τι αφορά το σύστημα αυτό υποχρεωτικής κατανομής θα πρέπει να τίθεται σε παραγωγή σε περιόδους κρίσης. Πώς ορίζεται όμως η περίοδος κρίσης από την Επιτροπή. Ενδεχομένως την επόμενη φορά θα υπάρξει ένας τέτοιος ορισμός. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, αν αναφέρονται τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης, ο σεβασμός των κριτηρίων αυτό είναι ένα στόχος για τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τα όσα ορίζονται από τις από Έθνη σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να υπάρξουν κριτήρια παρεφερή με αυτά του, ε, της Κοπεχάγης. Η Σιλβί Γκυγιόμ. Ευχαριστώ. Το θέμα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Ασφαλών Χωρών είναι παλιό, το είχαμε συζητήσει και το 2013 για την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τις διαδικασίες του, ότι είχαμε καταργήσει την, τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ασφαλών Χωρών για εθνικούς, αλλά ήταν μια ρεαλιστική επιλογή. Η οδηγία περιλαμβάνει ωστόσο σημαντικά πλαίσια για να διευκολύνει μια διατύπωση αυτού του καταλόγου από την Επιτροπή. Υπάρχουν διευκρινήσει για το πώς διαμορφώνονται οι λίστες, πώς, τι, τι λαμβάνουμε υπόψη και τρόποι καθώς και επιπλέον εγγύησει για τους ενδιαφερόμενους. Το λέω αυτό διότι στην πρόταση της Επιτροπής γίνεται μνήα για, σεβασμό, για το σεβασμό των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην οδηγία, ιδίω ό,τι αφορά τις διαδικαστικές και δικονομικές εγγύησεις. Είναι αναγκαίο να διαπιστώσουμε ότι μετά την υιοθέτηση της οδηγίας αυτής που περιλαμβάνει τη ρητή μνήμα για την ασφαλή χώρα καταγωγής, η διαφορετική αντιμετώπιση σε πολλές χώρες και η αντιμετώπιση αυτής καθεαυτής αυτής της ενές δημιουργία ανισότητες μεταξύ των χωρών. Συμφωνώ με τις ανησυχίες για την χρήση ε, των κριτηρίων της Κοπενχάγης ε, σαν δεδομένων για τις ασφαλείς χώρες καταγωγής. Να προσθέσω επίσης για την Τουρκία, ιδίως, το είπαν και κάποιοι προηγουμένως, 25% είναι το ποσοστό αναγνώρισης αυτή τη στιγμή για Τούρκους. Επίσης για το πώς μια χώρα βγαίνει από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ασφαλών Χωρών Καταγωγής και πώς εφαρμόζεται τούτο σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, αν μια χώρα που είναι στον ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή λίστα αλλάζει για αλλαγή, λόγω αλλαγή κατάσταση, τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Αυτό, αυτές φεύγουν από τον εθνικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι αν γίνει το αντίστροφο, δηλαδή φύγει από τον ευρωπαϊκό κατάλογο, είναι υποχρεωτική η αφαίρεση της χώρας αυτής και από τους εθνικούς καταλόγους. Η κυρία Φελέρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά και θα ήθελα να αναφέρω αρκετά κάποια θέματα που με ενδιαφέρουν πολύ. Ε, τα έχουν δείξει κι άλλοι. Όσον αφορά τις ε, επιθυμίες ε, του ετούντος άσυλο, ε, σε σχέση με την κατάσταση. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι στο θέμα αυτό η Κομισιόν στηρίζει το Κοινοβούλιο. Δηλαδή λέει ότι πράγματι πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι επιθυμίες του ετούντος άσυλο ε, για να μην γίνεται εκ των υστέρων δεύτερη μετεγκατάσταση. Ε, το Συμβούλιο τοποθετήθηκε, η θέση του ήταν πιο αρνητική κατά κάποιον τρόπο εδώ μπορούμε να μιλάμε και για εκτοπισμό. Δηλαδή τους μεταφέρουν τους ετούντες άσυλου σε μια χώρα ή σε ένα σε μια περιοχή που δεν αισθάνονται καθόλου καλά. Και θέλω να ακούσω εδώ την άποψη της Επιτροπής. Τι πιστεύει η Επιτροπή. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι οι επιθυμίες του ετούντος άσυλο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, όσον αφορά τον κατάλογο των ασφαλών ε, χωρών, η κατάσταση είναι η εξής. Στην Τουρκία, ας πάρουμε την Τουρκία η ελευθεροτυπία, ε, δεν θα το έλεγε και ότι υπάρχει και ελευθεροτυπία στην Τουρκία, ούτε και, ε, και χειρία κατάπαυση πυρός. Η Κομισιόν λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ταχύτατες διαδικασίες και πώς θα γίνει αυτό. Μπαίνουν στην Τουρκία και τι εκεί θα γίνεται η εξέταση των αιτήσεων. Πώς το βλέπει αυτό η Κομισιόν. Μετά η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτούς που έχουν ε, διαφύγει από εμπόλυμη ε, ζώνη. Εδώ συμφωνώ. Εντάξει, αλλά τι θα κάνουμε με όλου του άλλου ε, που είναι πρόσφυγες, οι οποίοι όμως δεν έρχονται από εμπόλεμες περιοχές, αλλά από περιοχές που υπάρχουν συγκρούσεις, εστίες κρίσεις και αυτοί είναι πάρα πολλοί. Και για αυτούς θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις γιατί αυτοί δεν εμπίπτουν στο μηχανισμό μετεγκατάστασης, αλλά κάτι πρέπει να σκεφτούμε και για αυτούς. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξτάσουμε σχετικά με τους ε, ετούντες άσυλο. Η κυρία Ντάλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται και θα εστιάσω την προσοχή μου στο μηχανισμό μετεγκατάστασης. Αυτό που προτείνει η Κομισιόν πράγματι είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούμε να τα εξετάζουμε όλα αυτά εν κενό, αυτό ήδη αναφέρθηκε. Και όλα αυτά θα λειτουργήσουν μόνο αν κατορθώσουμε να τροποποιήσουμε το Δουβλίνο με έναν τρόπο ε, που θα βγάζει νόημα και που θα δίνει τη δυνατότητα να παράγει αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ και χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει η συνθήκη του Δουβλίνου και αυτές οι διάφορες λύσεις που προτείνονται είναι ελένδετες μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κάποια λύση που να μπορεί κανείς να εξτάσει μόνη της εν κενό όπως λέω, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του και τα συνεπακόλουθα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν όσον αφορά το μηχανισμό με την κατάσταση. Η Κομισιόν λέει ότι αυτός ο μηχανισμός ε, χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μήπως μπορεί η Κομισιόν να μας εξηγήσει περισσότερο τι είναι αυτό ακριβώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αφορά ένα μόνο κράτος μέλος. Και τα λέω όλα αυτά διότι κατά το παρελθόν είχαμε καταστάσεις όπου μία χώρα και αναφέρομαι εδώ στη Μάλτα ε, κατέφυγε σε κάποιο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης που αφορούσε όμως μόνο τη Μάλτα, όχι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι άλλο που έχει σχέση με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρεται ότι ο μηχανισμός βασίζεται σε τέσσερα κριτήρια πληθυσμός, ΑΕΠ, ανεργία και ε, άσυλο κατά κεφαλή. Δυστυχώς όμως η Κομισιόν δεν αναφέρει το μέγεθος του κράτους μέλους και θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή τους από αυτό. Διότι εγώ πιστεύω ότι το μέγεθος του κράτους και οι δυνατότητες αυτού είναι καθοριστική σημασία και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα κριτήρια. Η κυρία Σκα Κέλλερ, παρακαλώ. Εντάξει, κάθομαι σε λάθος θέση, αλλά μπας θα μιλήσω από εδώ. Ευχαριστώ. Το σημαντικότερο είναι να περάσει αυτός ο μόνιμος μηχανισμός μετεγκατάστασης. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα επίγον ζήτημα μετά το άλλο. σήμερα αυτή την εβδομάδα ξέρουμε τι γίνεται, αλλά δεν ξέρουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα μόνιμο πρόγραμμα για αντίστοιχε επίγουσες καταστάσει. Αυτό πρέπει να προέλθει από το Συμβούλιο. Και εμεί, ω Κοινοβούλιο θέλουμε ω κανονικοί συνομοθέτε να μετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ με του συναδέλφου που ανέφεραν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προτεραιότητε και οι ανάγκε των προσφύγων. Αλλιώ δεν θα, θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε δευτερογενεί μετακινήσει. Η κατασταλτική εξέγγιση που ακολουθεί το Συμβούλιο και η Κομισιόν πρόσφατα πάει λάθος, σε λάθος κατεύθυνση. Διότι ε, η παραβίαση των δικαιωμάτων των ετούντων, των προσφύγων, ακόμα και των αναγνωρισμένων, είναι εις βάρος τελικά και των δικών μας συμφερόντων. Πρέπει να ξέρουμε πρώτα τι θέλουμε να αλλάξουμε σε μόνιμη βάση, όχι μόνο επιγόντως. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι τα κατασταλτικά μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα των πολιτών, που είναι κανονικοί ετούντες και μετά κανονικοί αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, δεν οδηγούν πουθενά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι και το κράτος υποδοχής και ο πρόσφυγας θα κερδίσουν από την απόφαση αυτή. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση του πρόσφυγα για το που θέλει να πάει, όντας ανοιχτή και όντας ευπρόσδεκτοι ε, και ε, όντας ανοιχτή στο να δεχθούμε. Αν μια χώρα δεν θέλει τον πρόσφυγα δεν θα πάει εκεί ο πρόσφυγας. Πρέπει λοιπόν να τους προσφέρουν και κάποια δυνατότητα διευκόλυνσης της εισόδου τους, της ένταξής τους. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα έχουμε πει σχεδόν όλα οι συναδελφοί μου. Δύο ερωτήσει μόνο. Το ένα είναι για τα hot spots που είναι πάρα πολύ σημαντικά σε όλη τη διαδικασία καταγραφή και επεξεργασία των ε, προσφύγων. Ακούμε για τα hot spots, αλλά ακόμα τουλάχιστον στη χώρα μου δεν τα έχουμε δει, δεν ξέρουμε πού βρίσκονται και θα θέλαμε την Κομίσιο να μα ενημερώσει για αυτά. Και το δεύτερο είναι με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε, μιλάμε για τον ε, πρόχειρο μηχανισμό, για τον έκτακτο και μιλάμε και για τον που ο έκτακτος είναι ήδη ξεπερασμένος ε, σε αριθμούς. Ε, τι θα τι βλέπει η Κομισιόν να γίνει όταν κάποιες χώρες αρνηθούν να πάρουν μέρος σε αυτόν τον έκτακτο, πόσο μάλλον στο μόνιμο μηχανισμό. Ποιες είναι οι εναλλακτικέ ιδέες που έχει. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Okay, um, ναι. Ευχαριστώ κύριε Κύρκο. Ο κύριος Χαραχάχο. Θα μιλήσω φιλανδικά. Η ερώτησή μου αφορά τον ορισμό των ασφαλών χωρών καταγωγής. Πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να συμφωνήσει σε μια κοινή προσέγγιση για χώρες όπως το Ιράκ, η Σομαλία ή οι περιοχές κοντά σε αυτές. Η ερμηνεία που ακολουθούν αυτή τη στιγμή τα κράτη για τις χώρες αυτές είναι ποικίλη. Κάποιες χώρες θεωρούν ότι κάποιες περιοχές του Ιράκ και της Σομαλίας είναι ασφαλείς. Δεν δέχονται ετούντες, από, δεν δέχονται πρόσφυγες από εκεί. Παρότι γενικά μπορεί τα άτομα αυτά να αξίζουν προστασίας. Χιλιάδες Ιρακινοί ταξίδεψαν μέχρι τη Φιλανδία μέσω Γερμανίας, Φιλανδίας, ε, Δανίας και Σουηδίας. Παρότι οι κανόνες λένε ότι θα πρέπει να ζητήσουν άσυλο στην πρώτη ασφαλή χώρα που πηγαίνουν. Αυτή η διαδικασία της αναζήτησης χώρας ασύλου θέτει σε κίνδυνο το σύστημα Σέγγεν, γιατί υποχρεώνει τα κράτη να αυξήσουν τους ελέγχους στα σύνορά τους. Αν δεν υπάρξει τέτοιος έλεγχος, θα υπάρξουν προβλήματα. The final, um... Ε, τελευταίος ομιλητής και η κυρία Χολμάγερ που ήρθε αργότερα δεν, είχε το χρόνο να μιλήσει ε, ως συντονίστρια. Οι υπόλοιποι θα μιλήσετε στον επόμενο γύρο. Έχουμε άλλα δύο τμήματα στη συζήτηση. Παρακαλώ να πειθαρχήσετε με την πρότασή μου. Τελευταίος ο μιλητής ο κύριος Ντεπρέ. Ζεράρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δική μου παρέμβαση είναι σε συνέχεια της παρέμβασης της Σεσίλια, την οποία προσυπογράφω. Άκουσα ότι πέθανε το Δουβλίνο, αυτή η πρώτη μου σκέψη σύμφωνα με το μηχανισμό που θέτουμε τώρα σε εφαρμογή. Αν το διαβάσουμε καλά θα δούμε ότι το 40% ε, των ατόμων που θα φτάσουν θα μπορούσαν να εντοπιστούν. Δηλαδή θα, μείνουν, ε, θα ασχοληθεί με αυτούς η χώρα υποδοχής. Υπάρχουν 200.000 ψήφοι που θα φτάσουν στην Ιταλία, αυτοί που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και 100.000 με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούν οι Ιταλικές αρχές. Για αυτό το μηχανισμό μιλάμε. Βεβαίως η αλληλεγγύη, είναι μια αλληλεγγύη κατά 40%. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να αποφύγουμε σλιδισμούς βεβαίως, δεν απαλλάσσουμε τις χώρες ε, από την ευθύνη που έχουν, αλλά θα δούμε τι σημαίνει στο ίμιση των χωρών. Δεύτερος, αυτό που λέει η Επιτροπή, δεν μπορεί να γίνει μετεγκατάσταση αν δεν ανήκουν σε μια εθνικότητα όπου το 75% αυτών που ζήτησαν να τύχουν των διατάξεων αυτών θεωρήθηκαν ότι θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί. Ποιες χώρες αφορά αυτό. Ε, εδώ αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες εθνικότητες που είναι επιλέξιμες συμφωνώ με την ύπαρξη ενός συστήματος ασφαλών χωρών καταγωγής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτές που συμπεριλαμβάνουν στους καταλόγους. Μία μόνο χώρα, η Τουρκία. Για ρίξτε μια ματιά, δέξτε πόσες αιτήσει γίνονται δεκτές για το φύρο 0,9%, Κόσοβο, Παυροβούνη, Σερβία. 24% όμως για την Τουρκία σε αντίθεση με όλα αυτά. Πέστε μου όμως, στην Τουρκία, επικεφαλής της Τουρκίας, βρίσκεται ένας πολεμοχαρής μεγαλομανής, ο οποίος στην ουσία έχει κηρύξει τον πόλεμο στον ίδιο το λαό του. Και μου φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό το να τα λέμε αυτά εδώ. Ένα άλλο ερώτημα στην Επιτροπή. Θα πρέπει να μεταφέρονται ε, οι άνθρωποι στις χώρες μετεγκατάστασης τι είδου έγγραφα θα πρέπει να έχουν, ποιο θα τα χορηγήσει αυτά τα ε, έγγραφα, τι θα είναι μια μεταβατική θεώρηση, ε, ποιο θα ορίσει αυτά τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη διέλευση των σύνορων. Τώρα, αυτά ε, που λέει η Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά διεξοδικότερα. Η Επιτροπή αξιολογεί όλα τα στοιχεία που βρίσκονται εδώ με κατεξιουδότηση ε, πράξη. Και μου φαίνεται ότι είναι ένα προνόμιο του εκτελεστικού που είναι ένα αρκετά σημαντικό. Κύριε Χολμάγερ. Κυρία Χολμάγερ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα όσον αφορά στο μηχανισμό μετεγκατάστασης, έχω τις εξής ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσει για το τι γίνεται με ένα κράτος από το οποίο κάποιοι μετανάστες αφαιρούνται για να μετεγκατασταθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Πώς ακριβώς γίνεται αυτή η κατανομή, γιατί μπορεί να αρχίσουν να τσακώνονται τα κράτη-μέλη. Ε, μπορεί κάποιοι να αναγκαστούν να πάρουν περισσότερους ε, από άλλους. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην προκύψουν αυτές οι έρηδες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το δεύτερο ερώτημα μου έχει, να κάνει, έχει σχέση με την ε, δυνατότητα κατάσταση ή τη μετεγκατάσταση ενός ε, ετούντος άσυλο ε, σε μια χώρα που δεν είναι όμως η χώρα η αγαπημένη του, η χώρα της επιλογής του. Τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή η Κομισιόν ε, θα επιτρέπει ή θα εμποδίζει τον ετούντο άσυλο να πηγαίνει σε αυτή τη χώρα. Γιατί τι νόημα έχει αυτός ο μηχανισμός αν ο τον άσυλο αποφασίζει μόνος του την επόμενη μέρα να πάει και που θέλει. Κάτι άλλο. Όσοι ζητάνε άσυλο. Κοιτάξτε, σε ορισμένα κράτη-μέλη, κυρίως στη Σουηδία και τη Γερμανία, το 1 τρίτο των, αρθόμων που, των ατόμων που καταφτάνουν δεν ετούνται άσυλο. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Όλοι αυτοί που έρχονται σε μας Πώς μπορούμε να τους επαναπροωθήσουμε χωρίς να αισθάνονται ότι είναι προσβεβλημένοι. Γιατί υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη μορφή αιτήσεως ασύλου. Υπάρχουν οι πρόσφυγες που λένε ότι δεν επιθυμούν δεν και δεν θέλουν να αιτηθούν ασύλο ούτε εδώ ούτε εκεί. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που ε, δεν είναι ετούντες άσυλο, σας λέω δεν θέλουν όλοι άσυλο, υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν. Τώρα, κάτι άλλο, όσον αφορά την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλησε το 24% τουλάχιστον ε, αυτό διάβασα σε αριθμούς που έχει υποβάλει η Γερμανία και διαπιστώνω ότι χορηγείται και δευτερογενής ε, προστασία διότι πολλοί έρχονται από τις ε, παραμεθόριες περιοχές με τη Συρία ή από εστίες κρίσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά την Τουρκία θα πρέπει να γίνεται αυστηρή ανάλυση των αριθμών για να γνωρίζουμε ακριβώς που υφίστανται τα προβλήματα. Και επίσης ε, για να καταλήξουμε τελικά αν θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους και εξετάζοντας το θέμα των Κούρδων της αντιμετώπισης των Κούρδων. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί με την Τουρκία ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που θα διεξάγουμε με αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Στίβενς. Ik Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Το νέο υποχρεωτικό πρόγραμμα δεν είναι επαρκές. Η Ευρώπη συνεχίζει να παραμένει θύμα των εθνικών πολιτικών. μας εκπλήσει αυτή η έλλειψη φιλοδοξιών. Από τη μία πλευρά υπάρχει αυτή η ροή προς την Ευρώπη με ένα δυσανάλογο αριθμό ετούντων άσυλο ενώ παράλληλα δεν υπάρχει μια σωστή εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων κανόνων, μολονότι βελτιώνονται οι διαδικασίες. Παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Ακόμα και τα αποκαλούμενα hot spots στα οποία θα έπρεπε να παρεμβαίνει η Frontex στην ουσία αμβλύνονται. Μία αλλαγή των υπαρχών των κανόνων. Δεν ξέρω που θα μπορούσε να οδηγήσει ελπίζω στο εσωτερικό του Συμβουλίου Υπουργών να υπάρξει ένα σύστημα που να λαμβάνει περισσότερο ε, υπόψη τα όσα αναφέρονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι με βρίσκει σύμφωνη το πρόγραμμα της Επιτροπής για μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ελπίζω να το έχουμε σύντομα. Μερικές ερωτήσεις για την Επιτροπή. Σχετικ... Πώς θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει ο καταμερισμός ευθυνών μεταξύ των χωρών μελών που μετεγκαθιστούν και αυτούς που υποδέχονται. Ποιος αποφασίζει, πόσα άτομα, ποιοι επιλέγονται, ποιος παίρνει την τελική απόφαση και πώς αυτό εφαρμόζεται πρακτικά λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό ατόμων που εισραίουν. Το άλλο ερώτημα αφορά τα παιδιά. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα μεταγκατάστασης για τα παιδιά ή για τους ε, ασυνόδευτους ανηλίκους ή για την επανένωση των οικογενειών. Τρίτον, προτείνατε να επανεργοποιήσετε την κατεξουσιοδότηση πράξη. Μπορείτε παρακαλώ να μας εξηγήσετε πώς έχει η κατάσταση, ποια είναι τα κριτήρια, πότε θα θεωρείτε ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η επόμενη ερώτησή μου είναι παρεφερής με αυτή που έθεσε η Μόνικα. Τι συμβαίνει αν κάποιος μετεγκατασταθεί σε μία χώρα μέλος. Αυτή η μετεγκατάσταση ισχύει μόνο για αυτή την ε, χώρα μέλος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικές χώρες που είναι περισσότερο ελκυστικές. Αν μετεγκατασταθεί σημαίνει ότι πάει κανείς σε μία χώρα μέλος και μετά πηγαίνει σε κάποια άλλη... Το πρόγραμμα, το, το, το πρόγραμμα αυτό καταραίει και βεβαίως τα πλαίσια της ε, απόλυτου, απόλυτου σεβασμού της ελευθερίας ε, επιλογής θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πραγματικός μηχανισμός μετεγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, έχω μια ερώτηση. Γιατί η Επιτροπή δεν ε, προτείνει ένα σύστημα επανεγκατάστασης αυτό ανοίγει περισσότερους δρόμους ε, νομικούς, γιατί δεν χρησιμοποιούμε την επανεγκατάσταση αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να διατρέξουν κινδύνους και να ταξιδεύσουν σε μια χώρα με εξωτερικά ε, σύνορα. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί εδώ. Ε, θα ήθελα να το εξηγήσει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφαλούς χώρας. Με βρίσκει σύμφωνη αυτή η πρόταση είναι κάπως περίεργο για μένα. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι θέμα αξιολόγησης. Όλη η συζήτηση γίνεται μια συζήτηση για την Τουρκία και εδώ μιλάμε για ατομική αξιολόγηση. Δεν θα σταλθούν ε, όλοι μαζί πάλι ε, στη, πίσω στην Τουρκία. Μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει χώρα μέλος που έχει το δικό της κατάλογο που είναι διαφορετικός από αυτόν που προτείνει η Επιτροπή. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι μπορεί να γίνει πρακτικά. Και το τρίτο ερώτημα. Τι θα συμβεί με την Γάμπια, το, την το Πακιστάν ή άλλες χώρες που έχουν οικονομικούς μετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες Βεβαίως ο καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο. Η Επιτροπή θα περιορίσει τον κατάλογο ασφαλών χωρών μόνο στις υποψήσεις χώρες ή θα, απασχολεί, θα σας απασχολήσουν και άλλες χώρες που υπάρχουν περισσότερο οικονομικοί μετανάστες παρά πρόσφυγες. Ο κύριος Κριέζη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνοπτικά θα μιλήσω γιατί πολλά τα είπαν ήδη άλλοι συνάδελφοι. Συμφωνώ με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο δεύτερο πακέτο μετανάστευσης από πλευράς Επιτροπής. Εύχομαι το Συμβούλιο να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και να ε, κάνει ένα μεγάλο βήμα μπρος σε στιγμές ιδίως όπου εντοπίζουμε κανόνες για τον μηχανισμό μόνιμης μετεγκατάστασης που είναι αρκετά ισορροπημένες. Ίσως το ποσοστό ανεργίας ε, με που υπολογίζεται μόνο στο 10% θα μπορούσε να αναθεωρηθεί, αλλά αυτό είναι λεπτομέρειε. Μια ερώτηση θέλω να θέσω για τον κατάλογο των ασφαλών χωρών καταγωγή. Εκεί όπου αναφέρθηκε ότι αν ο ετών είναι πολίτη ενό των κρατών που περιλαμβάνει ο κατάλογος αυτό, το αίτημα εξετάζεται παρά τα αυτά. Τι πλονεκτήματα υπάρχουν σε εισαγωγικά τα πλονεκτήματα ως προς την ταχύτητα της εξέτασης του αιτήματος. Τι περιλαμβάνει είναι αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο θέμα του επαναπατρισμού, της επιστροφής όσων δεν δικαιούνται πολιτικού ασύλου ή άλλου είδους διεθνούς προστασίας. Αυτό που έγινε το 2013 είναι ενδεικτικό κάτω από 40% αυτών που έπρεπε να επαναπατριστούν, πρίστηκαν ουσιαστικά. Η Ευρώπη πρέπει και στο σημείο αυτό να κάνει περισσότερο, διακρίνοντας καλύτερα μεταξύ ετούντων των προσφύγων και αυτών που έχουν οικονομικό, αυτών που μετακινούνται για οικονομικούς λόγους. Οι δύο εισηγητές τώρα, για την ολιστική προσέγγιση θέλετε να μιλήσετε, δεν λείπατε στο ξεκίνημα συνάδελφοι. Ή θέλετε να μιλήσετε για τα επόμενα δύο ζητήματα, ίσως να θέλετε να συνοψίσετε. Πιστεύω ότι τα επόμενα δύο θέματα θα είναι πιο σύντομα. Θέλετε τώρα να μιλήσετε στο τέλος της συζήτηση. Τώρα θέλετε να μιλήσετε. Ναι, τώρα. Οπότε μιλήστε. Πρόεδρε, μετά πρέπει να φύγω, γι' αυτό θέλω να μιλήσω τώρα. Κάποιε παρατηρήσει. κάποιες παρατηρήσεις. Είναι θετικό το ότι το συζητήσαμε το θέμα αυτό σήμερα, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών. Οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας υποβάλλονται υπό τη μορφή της συναπόφασης Δηλαδή είμαστε στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο. Αυτό είναι θετικό. Θα ξέρουμε περισσότερο το απόγευμα, αλλά πιστεύω ότι την θέση μας εδώ πρέπει να την κρατήσουμε. Ελπίζω απόψε να μην έχουμε τα ίδια με την περασμένη εβδομάδα. Κράτη-μέλη να επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους και να μην ε, ε, αλλάζουν γνώμη και αυτό να φτάσει μέχρι ε, τη σύνοδο κορυφής. Για τη μετεγκατάσταση πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδούμε τα κριτήρια ούτως ώστε να μην έχουμε ένα μηχανισμό που θα είναι δυσανάλογο για την α ή τη β χώρα. Το βασικό μου θέμα είναι η πρόταση αυτή να γίνει δεκτή, γιατί πάντα περιμέναμε, μας λέγανε μάλλον ότι η προσωρινή η νομοθεσία την προσωρινή προστασία δεν μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί λόγω των ε, προς κομμάτων της Επιτροπής. Ελπίζω να υπάρχει ένας οργανισμός που θα λειτουργήσει. Σε ό,τι αφορά τις ατομικές προτιμήσεις, πολλοί είπαν ότι δεν συμφωνούν και επιμένουν ε, να λαμβάνονται υπόψη προτιμήσεις των προς μετεγκατάσταση ετούντων. Εμείς συμφωνούμε. Στο ψήφισμα που εγκρίναμε πριν από δύο εβδομάδες, το είπαμε. ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνει η διαδικασία, να λαμβάνει υπόψη την, τα δικαιώματα των προσφύγων και μάλιστα να είναι στο κέντρο των δρασεών μας. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό ως δικαιολογία για να μην δέχονται άτομα και να λένε «Μα δεν θέλει κανείς να έρθει στη χώρα μας, και γι' αυτό να μην παρέχουν ένα ενδεδειγμένο σύστημα ασύλου. Θα πρέπει να υπάρξει μια πίεση από πλευρά μα για τον κατάλογο των τρίτων των ασφαλών χωρών καταγωγή είναι κάτι που η ομάδα μου πάντα ζητούσε. Αν δούμε τις εκθέσεις του ΕΑΖΟ θα διαπιστώσουμε τεράστιες αποκλήσει μεταξύ κρατών μελών ως προς το πώς εξετάζουν τις διάφορες χώρες με βάση τις σχέσεις τους με τις συγκεκριμένες χώρες. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που αναφέρουν ότι πρέπει να ξέρουμε περισσότερα. Αν θα υπάρξει περισσότερη συζήτηση για τις χώρες καταγωγής, σε περίπτωση ιδίω που τα άτομα που έρχονται στην χώρα μας δεν δικαιούνται προστασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα προτιμούσα να πάρω το λόγο αφού μιλήσουμε για τα δύο επόμενα σημεία. Όλα. Να περάσουμε τώρα δίνοντα το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, υποβλήθηκαν περίπου 80 80 ερωτήσεις στην Επιτροπή. Κοιτάξτε, υπάρχουν και υποερωτήσεις ε, για να είμαστε έτσι δίκαιοι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω στις περισσότερες εξ αυτών, αλλά υπάρχει και η νομοθετική πρόταση για τις ε, θεωρήσεις. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε αργότερα όταν θα εξετάσουμε τις ε, νομοθετικές προτάσεις στην Επιτροπή. Να σας πω και εγώ κάτι. Πράγματι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες και πολύ εξειδικευμένες ερωτήσεις που τέθησαν, ε, αλλά ε, απλά θέλω να το διευκρινίσω ότι υπάρχουν και πολλές και ουσιαστικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τα hot spots, ε, αυτά τα κέντρα καταγραφής, νομίζω είναι απόλυτα σαφές για όλους μας ότι πρέπει να έχουμε την πρωτοβουλία των αρμόδιων ε, φορέων τη ΕΑΖΟ, παραδείγματος χάνει και άλλων, για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα μετεγκατάσταση. Αυτό το κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Έχουμε αναπτύξει εκεί προσωπικό και επίση ε, έχουμε ε, συστήσει δύο περιφερικά γραφεία, το ένα στην Κατάνια και το άλλο στον Πειραιά, στην Ελλάδα, όπου συντονίζουμε τις ε, ενέργειες ε, των φορέων για να εφαρμόζεται το σύστημα, γίνεται η δακτυλοσκόπηση και μετά εφαρμόζεται η υπόλοιπη κοινωτική νομοθεσία. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία κλειδί και έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα στο θέμα του Δουβλίνου, το αν έχει πεθάνει ή όχι το Δουβλίνο, ε, φιλοσοφικό το ερώτημα, αλλά στην πραγματικότητα το Δουβλίνο δεν έχει πεθάνει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τροποποιήσουμε τη συμφωνία του Δουβλίνου, να συνδέσουμε τη συμφωνία αυτή με ένα μόνιμο μηχανισμό έτσι ώστε να βελτιωθεί αυτό το σύστημα του Δουβλίνου. Πάντως η αρχή, σε επίπεδο αρχής, το να μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στις ε, χώρες από τις οποίες εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η αρχή παραμένει. Ε, το μόνο που κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε ένα σύστημα που να βοηθάει τις χώρες λόγω της συμφωνίας του Ντουβλίνου. Αλλά κατά τα άλλα η συμφωνία του Ντουβλίνου πρέπει να παραμείνει. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν που θέλουν να πάνε. Αυτοί φεύγουν ε, γιατί φοβούνται για τη ζωή τους αλλά το να είναι κανείς ετών άσυλο δεν μπορεί να επιλέγει να πάει οπωσδήποτε στη Γερμανία ή στη Σουηδία αυτό εξάλλουν και το μήνυμα του μηχανισμού μετεγκατάστασης Τώρα, ε, εάν επιτρέψουμε τη δεύτερη μετακίνηση, τότε πια δεν λειτουργεί το σύστημα μεταγκατάστασης και δεν λειτουργεί και η Συμφωνία του Δουβλίνου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, δευτερογενείς μετακινήσεις θα περιορίζονται ε, στο βαθμό του δυνατού. Τώρα, ορισμένα μέλη λένε ότι οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν. Όχι δεν μπορούν να επιλέξουν, δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη χώρα που θέλουν να πάνε, ε, γιατί αλλιώ θα δείτε όλοι θα πάνε είτε στη Γερμανία είτε στη Σουηδία. Και δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι δίκαιη ε, απάντηση στα ερωτήματα που τίθενται. Άρα δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας τις προτιμήσεις των ετούντων άσυλων αλλά με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Ας πούμε το θέμα της γλώσσας. Αν κάποιος ετών πράγματι μιλάει γερμανικά εντάξει οτι είναι λογικό να πάει στη Γερμανία ή τα επαγγελματικά τους προσόντα. Με λίγα λόγια, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις προτιμήσεις τους, αλλά δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής της χώρας. Άρα δηλαδή αυτό πρέπει να το έχει κανείς κατά νου. Και τα κράτη-μέλη ε, και αυτά μετεγκαθιστούν τους ετούντες ε, μέσα στην ίδια τη χώρα λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις τους αλλά δεν υπάρχει η ε, εγγύηση ότι ο ετών θα πάει εκεί που θέλει. Όσον αφορά τώρα τις δευτερογενείς μετακινήσεις, αν κάποιος ας πούμε, πάει στην Πολωνία και μετά από δύο ε, μέρες βρεθεί στη Γερμανία, τότε πράγματι οι γερμανικές αρχές έχουν το δικαίωμα να τον επαναπροωθήσουν στην Πολωνία. Όσον αφορά τώρα στο δικαίωμα του ετούντος της ελεύθερης μετακίνησης, ο ετών μπορεί να μετακινείται μέσα στη ζώνη Σέγκεν, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος, τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε χρόνια. Άρα δηλαδή οι ετούντες, εντάξει μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στη ζώνη του Σέγκεν αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος, τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Όσον αφορά τον ΕΑΖΟ, ο ΕΑΖΟ δεν έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο, ε, βλέπετε υπάρχουν τα hot spot, τα σημεία καταγραφής, ο ΕΑΖΟ ε, συνεπικουρεί τα κράτη-μέλη για να επεξεργάζονται τις αιτήσει, ε, βοηθάει στο να καταγράφονται οι προτιμήσεις τους και πάρα πολλά άλλα, όμως ο ΕΑΖΟ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες ασύλου, ε, στις ε, χώρες όπου δέχονται μεγάλη πίεση. Για ένα πολύ απλό λόγο, ο οργανισμός αυτός έχει 80 άτομα. Ας μην ζητάμε λοιπόν υπερβολικά από ένα οργανισμό με 80 άτομα. Στη Γερμανία, ο γερμανικός οργανισμός ε, ασύλου τώρα τρέχει τη διαδικασία για να προσλάβει 2.000 άτομα. Έτσι λοιπόν, αν δεν αυξηθεί το προσωπικό του Άζο σε 20.000, δηλαδή τον αριθμό που έχουν τώρα επί χίλια, όσον αφορά το προσωπικό, αν δεν γίνει αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Απλά σας το επισημαίνω ότι πρέπει να είναι κανείς ε, λογικός όταν ζητάει από τη Frontex ή από τον ΕΑΖΟ να χειριστούν το θέμα της κρίσης. Όσον αφορά τώρα τις ε, τρίτες χώρες ως χώρες προέλευσης, ο κατάλογος που έχουμε καταθέσει δεν καλύπτει τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης δεν είναι προϋπόθεση για να τοποθετηθεί μια χώρα στον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Αυτός ο κατάλογος είναι στο, σε παράρτημα της οδηγίας που έχει εκδοθεί. Εμείς απλά χρησιμοποιούμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης και λέμε ότι οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να καλύπτουν τα κριτήρια της ε, Κοπενχάγης. Πάντως ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και όπως αναφέρεται και στο επεξηγηματικό παράτημα της πρότασης, ε, εμείς θέλουμε να εξετάσουμε και άλλες χώρες, χώρες της Αφρικής, να προσθετούν σε αυτόν τον κατάλογο περισσότερες χώρες. Για να γίνει όμως αυτό χρειαζόμαστε μια καλή ανάλυση της ε, ε, οποιασδήποτε χώρας ε, συζητάμε. Η Γκάμπια ας πούμε συζητήθηκε αλλά πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση στην Γκάμπια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και το καθεξής και προς το παρόν δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για τα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε στοιχεία γιατί συζητάμε ας πούμε για την ένταξή τους. Το κεφάλαιο 20 γίνεται ε, συζητήσεις ε, για θέματα σύλλου κράτους δικαίου. Άρα δηλαδή εκεί υπάρχει μόνιμη παρακολούθηση, ε, υποβάλλονται εκθέσεις και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μπορούμε να τις τοποθετήσουμε στον κατάλογο. Όπως πολύ σωστά ελέγχθη από πολλούς βουλευτές, ο κατάλογος αυτός δεν αποκλεί βέβαια ότι ε, θα λαμβάνονται υπόψη και με μονομένες περιπτώσεις. Και το να είναι κανείς στον κατάλογο αυτό απλά σημαίνει ότι μας δίνει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε επιταχυμένες διαδικασίες. Ένα ετών πάντα μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι η περίπτωση του, στη συγκεκριμένη περίπτωση του η Τουρκία δεν θα ήταν ε, ασφαλής χώρα. Ας μιλήσουμε λοιπόν πιο ανοιχτά. Ένας Κούρδος έρχεται και ζητά άσυλο στην Ελλάδα και μας λέει ότι δεν αισθάνεται ασφαλής στην Τουρκία, έχει δικαίωμα να λάβει προστασία στην Ευρώπη αν μπορεί να το αποδείξει. Δεν αποκλείει την χορήγηση ασύλου σε κάποιους, αλλά την, δεν το δεν αποκλείεται η προστασία τους, απλώς οι διαδικασίες είναι πιο γρήγορες και επιτρέπει στις υπηρεσίες να επικεντρώνουν ε, την προσοχή τους στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Πολλοί αναφέρθηκαν στους Ρωμά. Αν δείτε το ποσοστό αναγνώρισης Ρωμά στην Ευρώπη, το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό. Οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι κριτήριο χορήγησης ασύλου γιατί σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να δώσεις καθεστώς πρόσφυγα σε πάρα πολύ κόσμο, ανά τον κόσμο. Οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι όρος, δεν είναι παρικής όρος για να δοθεί άσυλο. Για τον κατάλογο αν μια χώρα φύγει από τον κατάλογο έχει επίπτωση στο, στον εθνικό κατάλογο, ναι. Θα συνεχίσει να υφίσταται ο εθνικός ε, κατάλογος, αν μια χώρα ωστόσο μπει στον ευρωπαϊκό κατάλογο, αναλαμβάνουμε εμείς. Η χώρα αυτή, ή ε, μάλλον η αντιμετώπιση της χώρας αυτής επιβάλλεται στα κράτη-μέλη. Ωστόσο, θέλουμε τη διατήρηση και των εθνικών καταλόγων, διότι κάποιες χώρες έχουν διαφορετικές ζωές ετούντων. Μπορεί να έχει περιπτώσεις όπου έχεις κάποιον από τον Μπάγκλαντες που ζητά άσυλο σε μία χώρα μόνο, όχι αλλού, μπορούν να το αντιμετωπίσουν ε, εθνικά. Με έλεγχο των εθνικών τους δικαστήριων. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο ωστόσο να είναι η συγκεκριμένη χώρα στον ευρωπαϊκό κατάλογο στη φάση αυτή. Μπορεί να συνεπάρξουν λοιπόν εθνική και ευρωπαϊκός κατάλογος. Να δω τι σημειώσεις μου μισό λεπτό. Για το 75% του κυρίου Ντεπρέ ήταν μια ερώτηση. Τι εννοούμε. Αν δείτε τις χώρες αυτή τη στιγμή που είναι πάνω από το 75% είναι η Συρία, η Ερυθρέα και το Ιράκ. Τρεις χώρες. Όταν εγκριθεί η πρόταση θα δούμε ποιες είναι οι χώρες που είναι πάνω από το 75%. Σε ένα χρόνο μπορεί οι χώρες να είναι διαφορετικές. Γιατί βάλαμε το όριο αυτό για να αποφύγουμε να υπάρχει μεγάλη μετακίνηση ατόμων μέσα στην Ένωση. Που δεν είναι σαφές ότι χρειάζονται διεθνή προστασία. Γιατί μπορεί να, να χρειάζεται να ληφθούν πολλές αποφάσεις επιστροφής, για παράδειγμα. Αν εφαρμόζεις το μηχανισμό ε, με την κατάσταση άτομα με χαμηλό ποσοστό ε, αναγνώρισης και φύγουν από την Ιταλία, την Ελλάδα στην Πολωνία μετά θα πρέπει να τον απορρίψουν οι Πολωνοί γιατί ε, το ποσοστό αναγνώρισης είναι χαμηλό τότε οι Πολωνοί θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία επιστροφής σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε ξοδέψει πολύ χρόνο και χρήμα και μετά πρέπει να προχωρήσουμε σε επιστροφή για τα host, η έννοια του hot είναι να επιτρέπουμε το γρηγότερο δυνατό την επιστροφή σε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας στο σημείο εισόδου στην Ευρώπη. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε άτομα με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας αποφεύγοντας την επανεγκατάστασή τους χωρίς πραγματικούς λόγους. Αυτό είναι το αίτιο του 75%. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ερώτηση γιατί όχι να, να, γιατί να έχουμε ένα μόνιμο πρόγραμμα επανεγκατάσταση. Σωστή ερώτηση. Ο πρόεδρος Γιόνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ανέφερε ότι του χρόνου θα υποβάλει η Επιτροπή ένα μόνιμο πρόγραμμα επανεγκατάστασης αναγνωρισμένων προσφύγων. και για λόγους ελεγγύης στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και για να αυξηθούν οι νομικοί δρόμοι εισόδου στην Ευρώπη. Αυτό που κάνουμε είναι το εξή. Χθε είχαμε μια συνάντηση με όλα τα κράτη-μέλη το και το ΕΑΖΟ για να συζητήσουμε τα πρακτικά θέματα εφαρμογή τους. Η διαδικασία είναι μια σύνθετη αν θέλετε. Μπορεί να έχουμε μια ειδική συνάντηση γι' αυτό. Η ιδέα είναι η Ιταλία και η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει υπόψη το προφίλ των ατόμων, να εντοπίσει αυτούς που είναι προς μετεγκατάσταση. Τα κράτη-μέλη θα έχουν στείλει μέσα σε ένα, σε τρεις μήνες τις ποσοστώσεις ή σε μια περίοδο δύο ετών ωστόσο. Η Φιλανδία παίρνει 2.000, θα πάρουν 500 του χρόνου, άλλους 500, του, τον άλλο μήνα, άλλους 500 αργότερα. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό έγκαιρα και μετά θα γίνει, αυτό γίνεται βάσει του αιτήματος των κρατών μελών. Μετά θα οριστούν τα άτομα προς μετεγκατάσταση, θα υπάρχουν έλεγχοι ασφάλειας, το ζήτημα του ποιες είναι αρχές που θα προχωρήσουν στην μετεγκατάσταση με την υποστήριξη δε, του ΔΟΜ, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, θα οργανώσουμε τη μεταφορά των ατόμων αυτών. Συνοπτικά αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Όπως είπα, ξεκινούμε με τις πρώτες 32.000 κάτι που νομίζω ανοίγει το δρόμο για το μόνιμο σύστημα με την κατάσταση που ελπίζουμε να εγκριθεί. Εμείς κρυκλούμε λοιπόν με τους 32.000, ελπίζουμε το απόγευμα να υπάρξει συμφωνία για τις 120.000 και θα έχουμε μια εμπειρία από αυτά τα δύο προσωρινά συστήματα με την κατάσταση που θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το μόνιμο σύστημα εντεγκαταστασης πολλα Πολλά κράτη-μέλη το είχαν τονίσει αυτό άλλωστε ότι χρειαζόμαστε ένα μόνιμο σύστημα και όχι να δουλεύουμε μόνο ad hoc. Ερέθησαν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το μηχανισμό κρίσης. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό στο κείμενο. Εμείς από τη σειρά μας είμαστε ανοιχτοί στο να υπάρξει ένας καλύτερος ορισμός. Εμείς λέμε ότι κρίση με τον όρο κρίση εννοούμε ε, μια κατάσταση που ασκεί πιέσεις ακόμα και σε ένα καλά προετοιμασμένο μηχανισμό ασύλου. Και θέλω να πω στην κυρία Μέσολα ότι λέει ο ορισμός λαμβάνοντας ε, υπόψη και την χώρα μέλος. Δεν είναι ένα κριτήριο που βασίζεται σε σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε τις πιέσεις που ασκούνται χώρα μέλος και λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος και την έκταση της χώρας μέλους. Σε ό,τι αφορά την κλίδα κατανομής και τα κριτήρια, ε, δεν βάλαμε το, την έκταση αλλά τον πληθυσμό της χώρας και, και τον αριθμό των ετούντων άσυλο κατά κεφαλή. Πιστεύουμε ότι ο πληθυσμός είναι σημαντικότερος από το, την έκταση της χώρας. Αλλά βεβαίως θα καταβάλουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την κλίδα κατανομής και να συζητήσουμε μαζί με το Κοινοβούλιο παράγοντες που αφορούν αυτή την, ε, το, τον τρόπο κατανομής. I think I will Κύριε Μισελ, αν κάποια χώρα μέλο θεωρεί ότι δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, ενδεχομένω θα μπορούσε να σας τις υποβάλει γραπτό. Μπορεί, μπορεί να σας υποβάλει γραπτός. Ε, μία, ένα από τα ερωτήματα αφορά τη μεταφορά από τη μία χώρα μέλος ε, στην άλλη. Χρησιμοποιείται ένα σύστημα λεσέ-πασέ, δηλαδή άδεια ε, διόδου. Μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα λεσέ-πασέ το οποίο προβλέπεται στη Συμφωνία του Δουβλίνου. Δεν είναι, δεν είναι μείζον θέμα πάντως. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σας περιμένει πολλή δουλειά. Κύριε Μισελ, νομίζω ότι δουλέψατε σκληρά σήμερα. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. της Εξωτερικής Υπηρεσίας δράση, σημείο 6 ως 10. Θέλετε να, τα... να μια ματιά σε αυτά και να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, προσπάθησα να καλύψω τέσσερα σημεία. Ενδεχομένω, μερικοί συνάδελφοι δεν ήταν εδώ από την ε, έναρξη της συζήτηση. Σας λέμε λοιπόν ότι την έχουμε διαρθρώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παρακαλώ κύριε Μισελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο σημείο αφορά την ανακοίνωση από την Επιτροπή σχετικά με τις ε, ε, προμήθειες, με τις δημόσιες συμβάσεις. η, ασκείται πιέσεις στις ε, δημόσιες αρχές και πολύ συχνά θα πρέπει να αυξήσουν τη δυνατότητα οι υποδοχής που έχουν να βρουν καταλήματα να διαπραγματευτούν ε, νέες συμβάσεις ε, για τροφοδοσίας, περίθαλψης κτλ. Εμείς θα θέλαμε να διευκολύνουμε τις δημόσιες συμβάσεις και τους κανόνες που τις διέπουν. Εδώ αναφέρουμε Ποιοι είναι οι υπάρχοντες κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα γρήγορο και άμεσα δυνάμενο να εφαρμοστεί τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μια νέα οδηγία ε, για τις δημόσιες συμβάσεις και αυτό θα εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να μπορούν να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Αυτό ό,τι αφορά το πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο για την, τον επαναπατρισμό. Για την, για την επιστροφή έχει υιοθετηθεί ένα νέο πακέτο για το θέμα της ε, επιστροφής. Εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία του συστήματος ε, αίτησης ασύλου. Αν το εξετάσουμε αυτό το ποσοστό επιστροφής, λέμε, βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δοκιμάζουν, απορρίπτονται και γνωρίζουν ότι η πιθανότητα επιστροφής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή το 40% των μεταναστών αυτών που εκλείσαν να φύγουν έφυγαν στην πραγματικότητα. Δηλαδή πάρα πολλοί δεν επιστρέφουν. Αυτό είναι ένα πολύ ε, προβληματικό σημείο γιατί στέλνει λάθος μηνύματα. Ανεπάρκειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης. Το προβληματικό θέμα της Επιτροπής, επιστροφής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ενδεχομένω χρειάζονται περισσότεροι πόροι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να υπάρξει επιστροφή σε χώρε που δεν συνεργάζονται. Προτείνουμε λοιπόν μία σειρά από για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος της Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την επιστροφή. Δεύτερον, επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την συνεργασία μας σε επίπεδο επανεισδοχής. Θα πρέπει να τονίσω ότι όλες οι δράσεις που προτείνουμε είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς συμβάσεις και συνάδρουμε και με τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Βεβαίως υπάρχει και η οδηγία επιστροφής που έχει πάρα, πολλά, ε, πάρα ε, ε, ρήτρε διασφάλιση, συνυπολογίζοντα βεβαίω το δικαίωμα που έχουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν. Σε επίπεδο νομοθεσίας θα ήθελα να πω ότι στο τέλος του χρόνου θα υποβάλουμε μία τροπολογία στον κανονισμό της Frontex για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εντολή της και προτείνουμε να υπάρξει, να δημιουργηθεί ένα γραφείο, ένα ειδικό γραφείο με ειδική υπηρεσία επιστροφής. Προτείνουμε και μερικές νομοθετικές τροπολογίες στο σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν για να το καταστήσουμε υποχρεωτικό. Από τη στιγμή δηλαδή που υπάρξει απόφαση επιστροφής θα πρέπει να είναι δυνατόν σε κάποιον να το εξετάσει, να το ελέγξει. Γιατί ε, Πολλέ φορέ γίνεται η άδεια για μία χώρα, η είσοδο γίνεται από τη μία άλλη και λοιπόν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Δύο νομοθετικέ προτάσεις. Επίσης αυξάνουμε τον προπολογισμό και την επάντρωση της Frontex για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις διαδικασίες επιστροφής. Αυτά όμως είναι θέματα που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκτενέστερα. ό,τι αφορά εξωτερικά θέματα. Θα θέλαμε να ενδυναμώσουμε συνεργασία μας με τις αφρικές χώρες, αφρικανικές χώρες, χώρες καταγωγής, εφαρμόζοντας τη συμφωνία που θα μπορούσε να είναι μια καλή βάση για τον επαναπατρισμό, για την επιστροφή. Προτείνουμε να ξεκινήσουν καινούργιες διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένες χώρες καταγωγής για να διευκολύνουμε την επανεισοχή. Βεβαίως, όταν μιλάμε για ασφαλείς χώρες, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη σωστή ενσωμάτωση των επαναπατρισσόμενων. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια χρηματοδότηση ενός προγράμματος ε, ε, επανένταξης. Ε, στην συνάντηση κορυφή, στην Βαλέτα μιλήσαμε για ένα ταμείο. Το άλλο φορά ένα εγχειρίδιο επαναπατρισμού. Εδώ υπάρχουν κατευθυντήριοι γραμμές, κατευθυντήριες οδηγίες ε, που αφορούν ε, τους φύλακες, τις ε, αρχές της αστυνομίας, τους υπεύθυνου για θέματα μετανάστευσης, για τους διάφορες φορείς παρακολούθησης και ελέγχου. Είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο που είναι παρεμφερές με αυτό του Σέγγεν είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό και άμεσα μπορεί να βοηθήσει τους άμεσα εμπλεκόμενους να αντιμετωπίσουν το θέματα που αφορούν την επιστροφή. Δεν δημιουργεί ε, μια καινούργια νομοθεσία είναι ένα θέμα καθαρά πρακτικό ένα κάτι που αφορά ε, ε, συμβάλλει στην επίλυση πρακτικών θεμάτων αυτό το εγχειρίδιο διαμορφώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια με βάση την οδηγία επιστροφής και η γραμματεία του Κοινοβουλίου επίσης συμμετείχε στη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου. Αυτά σε ό,τι αφορά την επιστροφή. Ε, ε, Τώρα, το Trust Fund για την Αφρική η κυρία Μογκερίνη είχε έφυγε στις 5 Σεπτεμβρίου σε μια μεικτή συνάντηση της ΑΦΕΤ, της ΛΥΜΠΕ και της ΔΕΒΕ και παρουσίασε κάπως ε, τις παραμέτρους αυτές. Όπως ξέρετε θα προχωρήσουμε για την σύνοδο της Βαλέτα το Νοέμβριο 11 και 12 ένα πακέτο κονδυλίων για το Trust Fund αυτό προς το παρόν μιλάμε για 1,8 δις ευρώ που θα αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη και μεταναστευτικού χαρακτήρα έργα για την ανάπτυξη μπορούν τα κράτη να συμβάλλουν περαιτέρω στο Trust Fund. Η ιδέα είναι να δώσουμε έμφαση σε έργα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, βοηθούν την ένταξη των μεταναστών, και αυξάνουν την ικανότητα υποδοχής στην Αφρική ατόμων που είναι διωγμένοι είτε πρόσφυγες είτε όχι βελτιώντας τις συνθήκες ε, διαβίωσής τους αλλά και έργα ανάπτυξης ε, αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Αφρική. Νομίζω ότι αυτά ήταν όλα. Ευχαριστώ συνάδελφοι, για το τμήμα αυτό θα ήθελα να μείνετε στο δίλεπτο παρεμβάσεων για να έρθει στις 11.30 προεδρία. Ξεκινούμε και πάλι με τους συντονιστές. Η κυρία Χολμάγερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ευχαριστώ καταρχάς την Επιτροπή για την εξαιρετικά λεπτομεριακή και σύντομη περιγραφή. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι όσον αφορά την επαναπρόσθεση δεν υπάρχει ε, νομοθετική πρόταση μέχρι στιγμή. Θα υπάρξει για να συζητήσουμε από αυτή. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ετούντων. Από την άλλη πλευρά να καταστεί σαφές ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει σε μία χώρα ε, θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον ε, ενδεχομένως να πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Γιατί αν δεν γίνει αυτή η επαναπρόθεση αυτό είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει κυρίως ε, την δυνατότητα άλλων που να έχουν αυτό το δικαίωμα. Ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μεγάλος αριθμός ετούντων άσυλο, ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές δαπάνες που δημιουργούνται. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τις τροποποίησεις στο σύστημα Schengen. Επίσης θα ήθελα όσον αφορά την επιστροφή, την επαναπρόθεση... Ε, να μας πει η Κομισιόν τι ακριβώς προτίθεται να κάνει πολύ συγκεκριμένα κατά τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και μήνες ε, για να έχουμε έτσι μια ιδέα το ε, κατά πόσον θα δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι θέλετε να αυξήσετε τον προπολογισμό και το, το προσωπικό της ΕΑΖΟ και της Frontex Εάν θελήσετε να βοηθήσετε τα κέντρα καταγραφής, ακόμα και στις περιπτώσεις επαναπρόθεσης, μπορείτε να μας πείτε λιγάκι τι έχετε κατά νου, τι αριθμούς προσωπικού θα θέλατε να υλοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω λέει κυρία Ζίπελ για αυτή την ε, ευθύνοπτη έκθεση της Επιτροπής. Όσον αφορά ε, τις ε, εντολές ε, που θα δίδονται. Νομίζω ότι πρέπει να δει κανεί κατά πόσο μπορούν να απλουστευτούν διαδικασίες. Όσον αφορά την επαναπρόθεση, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές ε, δεν γίνεται επαναπρόθεση για διάφορους λόγους. Υπάρχουν κράτη-μέλη που κατά το παρελθόν αυτό δεν το έβρισκαν σημαντικό γιατί δεν ήταν μεγάλη αριθμή. Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις όπου για ανθρωπιστικούς και πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επαναπρόθεση και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και εδώ θα ήθελα να τσω κάτι σε σχέση με το εγχειρίδιο. Πρέπει να σας πω ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες ε, απευθύνθηκαν ε, σε μένα ανήσυχοι πολίτες ε, που φοβούνται ότι η επαναπρόθεση θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με τη βία. Και νομίζω ότι θα πρέπει λιγάκι να το δούμε αυτό, κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και τι θα κάνουμε αν συμβεί όσον αφορά External Action και Trust Funds. Θέλω να σας επισημάνω ότι η χαρτική κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους απόλυτους αριθμούς των προσφύγων αλλά με την αδράνεια, τη μη πράξη των κρατών μελών. Και υπήρξαν κάποιες ε, υποσχέσεις ε, ότι θα εκταμιευτούν κάποια κονδύλια από την τη αρμοστία του προσφυγέ για πρόσφυγες αλλά δεν δόθηκε σχεδόν τίποτα. Τώρα για το Trust Fund και εγώ διαρωτώ πράγματι θα συμβάλλει αυτό το ταμείο έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη και εγκαταλείπουν την πατρίδα τους γιατί δεν έχουν καμία απόλυτη ελπίδα και είναι ακραίως φτωχοί αυτοί τι δικαιώματα έχουν. Βοηθούνται και τα χρήματα μήπως χρησιμοποιούνται απλά και μόνο για να γίνονται έλεγχοι τις ε, πατρίδες ε, των ανθρώπων αυτών. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό δεν καταπολεμούμε τα αίτια της ε, προσφυγιάς. Το ότι θα υπάρχει του χρόνου μία ακριβής μεταγκατάσταση, αυτό είναι σωστό. Όσον αφορά τα hot spot, θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Ανάμεσα στα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, πολλές και διαφορετικές ε, διαδικασίες ε, οι οποίες έχουν σχέση με τις οδηγίες περί ασύλου και πώς είναι δυνατόν σε ένα κέντρο καταγραφής ε, να αποφασίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα αυτός που είναι μπροστά μου είναι πρόσφυγας ή είναι κάποιος που πρέπει να γυρίσει πίσω. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται και η απόφαση που λαμβάνεται δεν θα πρέπει να εντάσσεται μέσα στη διαδικασία σύλλου. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί να πω ότι θα υπάρξει αύριο μια ειδική ακρόση ε, για τα hot spots, για τα κέντρα ε, καταγραφής. Λοιπόν, θα μιλήσω σου ειδικά. Γι' αυτό παρακαλώ να βάλετε όλοι τα ακουστικά σας. Και όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την παρουσίαση, για την ανακεφαλαίωση. Ε, τα ερωτήματά μας απαντήθηκαν, ίσως όχι πλήρως, αλλά τουλάχιστον ε, αναφέρθηκαν και νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι έχει κανείς τελικά το αίσθημα ότι μπορεί να συμβάλλει το να υπάρχει αυτό το ε, καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, αυτό είναι καλό για να μην ξεκινάνε καταρχήν οι άνθρωποι το ταξίδι. Επίσης, θα πρέπει να εξετάζουμε και την κατάσταση που υπάρχει. Για σκεφτείτε λιγάκι τους καταβλισμούς των προσφύγων. Εκεί λείπουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου χρήματα. Και γίνονται τα πάντα έτσι ώστε και η δουλειά να γίνεται κάπως ικανοποιητικά. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ φέρουμε πολύ μεγάλη ευθύνη η κατάσταση λοιπόν. Η Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ τα είπε πάρα πολύ καλά. Είπε ότι θα πρέπει να δούμε λιγάκι αυτό το θέμα της ε, ε, μετεγκατάστασης έτσι ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες ζωής. Και είναι ένα σκάνδαλο ότι μόνο το 15% των κρατών μελών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δέχονται τους πρόσφυγες με τη μετεγκατάσταση Άλλα 13 δεν δέχονται τίποτα. Και θέλω να σας πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εκείνη η χώρα του κόσμου που δέχεται τους περισσότερους. 70% και εμείς στο, στα 28 κρατημέλη δεχόμεθα μόνο το 12%. Αυτό λοιπόν είναι σκανδαλώδες, αν το δείτε πιο προσεκτικά. Σήμερα το πρωί Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων και που μπορούμε να δείξουμε και θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας για την ιδιαίτερα επικοδομητική αυτή συζήτηση. Παρακαλώ. Η Τζούντιθ είναι εδώ. Η Λόρα. Η κυρία Μέιερ. Όχι. Γιώτοβα. Κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Σας παρακαλώ να βάλετε τα ακουσικά σας. Δύο ερωτήσεις. Ο κανονισμός για τη Frontex θα κατευθυνθεί προς τα πού. Θα αφορά ένα φορέ παραπατρισμού. Ή θα ακολουθήσετε την άποψη ε, χωρών μελών που θέλουν να ενισχύσουν τα σύνορα, τα... τη φύλαξη των σύνορων. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν το στρατό για τη φύλαξη των συνόρων. Δεύτερη ερώτηση. Αυτά που προτείνατε και που συζητήσαμε τις τελευταίες πέντε μέρες αφορούν το προσωρινό μηχανισμό και το μόνιμο μηχανισμό. Υπάρχει, ε, σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει ένα πλαν B. Ο κύριος, ο Πίτερ Ντίτερ Πίτερ. Εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι για το τρίτο και τέταρτο σημείο της συζήτησης, αλλά νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Α, θα φύγετε. Για το τρία και το τέσσερα, μηχανισμό επανεγκατάστασης. Ωραία, πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το να βεβαιωθούμε να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε δύο σοβαρά προβλήματα με τον μηχανισμό επανεγκατάστασης και με τον κοινό κατάλογο. Ο μηχανισμός επανεγκατάστασης είναι μόνο το πρώτο βήμα και χρειαζόμαστε ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό ενσωμάτωσης των προσθήκων για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, άκουσα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να μιλάει για ένα κοινό κατάλογο, ευρωπαϊκό κατάλογο και ένα εθνικό κατάλογο. Βεβαίως στην περίπτωση της Ουγγαρίας βλέπουμε ότι στον εθνικό κατάλογο ασφαλών χωρών παίζονται διάφορα πολιτικά παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας κοινός ευρωπαϊκός κατάλογος ασφαλών χωρών διέλευσης και καταγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν Εθνική, αλλά να υπάρχει και ο ευρωπαϊκός. Ευχαριστώ. Επόμενος, Τσόμος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν διάβασα τα έγγραφα πρέπει να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα με τόσο φιλόδοξους στόχους ε, και χάρηκα που υπέβαλε και συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα, όσον αφορά τον κατάλογο των ασφαλών χωρών, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τον κατάλογο αυτό, Συμφωνώ και της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης, όμως θα ήθελα να προσθέσω και άλλες χώρες όπως το Μπαγκλαντές και η Σρι Λάνκα. Ο κατάλογος ε, των ασφαλών χωρών ε, για μένα αφορά και την Τινησία και την Αίγυπτο. Και θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οι πολίτες από αυτές τις χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ε, τώρα, ε, σχετικά με την επαναπρόθεση, η κυρία Χολμάια είπε ότι δεν αρκεί να απορρίπτεται η αίτηση, πρέπει πράγματι οι άνθρωποι αυτοί να επαναπροωθούνται. Πολλοί που έρχονται από τις αφρικανικές χώρες ε, έρχονται στην Ευρώπη και πρέπει να τους επαναπροωθήσουμε με ασφαλή τρόπο γιατί αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν στα χέρια εγκληματιών ε, τους χρησιμοποιούν ως σκλάβους. Αν λοιπόν αυτοί επαναπροωθηθούν ε, στη Λιβύη θα συμβεί αυτό που έγινε στους καταβλισμούς στη Σικελία. Δηλαδή έρχονται σε επαφή με ανθρώπους αυτούς και τους χρησιμοποιούν οι διακινητές ως σκλάβους. Αυτό πρέπει να το εμποδίσουμε. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και μπορεί να προσπαθήσει να συμφωνήσει με τις αφρικανικές χώρες για το κάτω από ποιες συνθήκες οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να επαναπροωθούνται. Παραδείγματος χάρη, στην Ιγυρία η παράνομη διακίνηση ανθρώπινων όντων είναι αξιόπινη πράξη, ε, κακούργημα που πολλές φορές όμως ε, δυστυχώς ε, δεν καταδικάζονται οι υποπτοί. Τώρα, όσον αφορά τις προθεσμίες ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική οδό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 Och det strömmar inte migranter till Europa. Det är väl inte... Πρέπει να μας εκπλήσει ιδιαίτερα αυτό. Γιατί ανοίγουμε τα σύνορά μας και εισραίουν ε, ομάδες μεταναστών. Στη Σουηδία υπάρχουν πολλοί που ζουν παράνομα και η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα του συλλάβει για να του στείλει και πάλι πίσω στη χώρα τους. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς ανοίξαμε ορθά τα σύνορά μας. Θα πρέπει λοιπόν να επαναφέρουμε τους ελέγχους στα σύνορα. Αυτό είναι κάτι που κάνουν πολλές χώρες μέλη. Σε ό,τι αφορά τους ετούντες άσυλο, μετά από 18 μήνες τα δακτυλικά αποτυπώματα διαγράφονται. Μπορούν λοιπόν να πάνε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκινήσουν και πάλι από την αρχή. ομάδες ολόκληρες μεταναστών που φτάνουν και κανένα δεν επιστρέφει στη χώρα του. Η κατάσταση έχει τεθεί εκτός ελέγχου. Υπόθηκε και προηγουμένως ε, ότι ματώνουν, ματώνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν έχουν πλέον χρήματα, δεν έχουν ε, ε, τρόφιμα για τους χιλιάδες ε, μετανάστες. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε εκεί που είναι, στη Συρία. Θα πρέπει να τους δώσουμε ε, πόσιμο... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βόιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, μιλήσατε πάρα πολύ σωστά για το θέμα της επαναπρόθεσης, αλλά ε, παραμένουν αρκετά σημεία διευκρινιστά. 40% πρέπει να επιστρέψουν ή επέστρεψαν και 60% παρέμειναν. Λέτε είναι Ιρακινοί. Τώρα τι είναι αυτά, είναι μέσος όρος ή είναι γενικά ποσοστά του συνόλου των μεταναστών που πρέπει να επιστρέψουν ή μήπω υπάρχουν ε, διαφορές ε, σε σχέση ε, όσον αφορά αυτούς που έρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια και αυτοί που κάνουν ψευδείς δηλώσεις. Γιατί ακούω όλο και περισσότεροι λένε ότι είναι σειροί γιατί υπάρχουν πολλοί, καταστρέφουν τα χαρτιά τους, λένε είναι Συρίοι, γίνονται δεκτοί ανεξάρτητα από το που έρχονται. Είπατε ότι η Frontex ε, ανοίγει ένα γραφείο επαναπρόθεσης με 81 υπαλλήλου. Πώς θα τα καταφέρατε, είπατε ότι θα αυξηθεί το προσωπικό. Στη Γερμανία, ας πούμε, πρόκειται να προσληφθούν 2.000 νέοι υπάλληλοι, Άρα εσείς ε, θα πρέπει να προσλάβετε 8.000 υπαλλήλους. Αυτά όμως όλα είναι μέτρα που αφορούν στην επαναπρόθεση, μέτρα όμως που δεν μπορούν να εφαρμοστούν όσο δεν υπάρχουν κίνητρα για τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και νομίζω ότι αυτό το καταπίστευμα δίνει μία δυνατότητα, αλλά πολύ περιορισμένη, ε, διότι βλέπουμε ότι ας πούμε ένας ε, ε, αυτών ε, θα χρηματοδοτείται με 5.000 ευρώ από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πατρίδα του για να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα να επιστρέψει ο άνθρωπος αυτός. Και όπως αναφέρθηκε ε, πολύ σωστά, οι άνθρωποι αυτοί ή μετακινούνται σε άλλη χώρα ή συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα κατά κόρον, δεν καταγράφονται καθόλου και αν δεν είναι κανείς ε, καταγεγραμμένος δεν μπορεί και να ε, επιστραφεί, να επαναπροωθηθεί πίσω στην πατρίδα του. Ο τελευταίος ομιλητής αυτή τη συζήτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά βάση χαιρετίζω την πρόταση της ε, Επιτροπής. Αυτά που παραθέτει είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει όμως να πω ότι είναι τραγικό ότι βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε γιατί είναι απόλυτα σαφές ότι τα βήματα και τα μέτρα που προτάθηκαν μολονότι είναι σωστά, έρχονται πάρα πολύ αργά και είναι ανεπαρκή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος όμως ε, να το συζητάμε τώρα. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να έχουν γίνει αυτά πριν από 5, πριν από 10 χρόνια. Ναι, χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικές ε, πολιτικές επιστροφής, χρειαζόμαστε σαφώς περισσότερους πόρους σε κάθε χώρα Ναι, θα χρειαστούμε έναν κοινό κατάλογο χωρών επιστροφής, αλλά Είναι λυπηρό το να διαπιστώνει κανείς ότι δεν υπάρχει ένα κοινό όραμα, μια κοινή άποψη για το πώς θα πρέπει να τα χειριστούμε όλα αυτά. Δεν κατηγορώ την Επιτροπή για το ότι έκανε πολύ λίγα και πολύ αργά, γιατί οι χώρες μέλη το βροντοφωνάζουν αλλά και κατηγορούνται αμοιβαίως ότι έγιναν πάρα πολύ λίγα. Ποιος φταίει για όλα αυτά, φταίνει οι κυβερνήσεις φταίνε για την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε τώρα. Δηλαδή γινόμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης που έχει τεθεί εκτός ελέγχου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει έλλειψη μιας κοινή αντιμετώπισης. Θα ήθελα να πω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής, όπως είπα, είναι προτάσεις που χρειαζόμαστε. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, Αλλά θερμή παράκληση. Ας το κάνουμε τώρα, αμέσως, γιατί ήδη, ήδη έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Ευχαριστώ. Πολύς χρόνος. Πάρα πολύς χρόνος. Μία σύντομη ερώτηση. Θα θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές και να διατυπώσω ένα σύντομο ερώτημα. Ο κύριος Σίπονα αναφέρθηκε σε αυτό το εγχειρίδιο η, επιστροφή, η Επιτροπή θα ήθελα να τους ευχαριστήσει για τη θαυμάσια δουλειά που έκαναν στον τόσο ευαίσθητο αυτό το τομέα. Η κυρία Σίπολ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Βεβαίως αυτά προσφέρθηκαν για πολλές ερμηνείες. Εγώ θα σας έλεγα να περιοριστούμε σε αυτό το θέμα, ε, το θέμα της κράτησης ας πούμε, τα ε, όρια της κράτησης. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θέματα λοιπόν που αφορούν την κράτηση. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθούμε και πάλι στο θέμα αυτού του εγχειριδίου, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Συνάδελφοι, θα έλεγα να περάσουμε στο σημείο 11 για τον χώρο του Σέγγεν. Μόλις η Επιτροπή θα συζητήσει αυτά τα θέματα. Εμεί θα προσεγγίσουμε τι 11 και 30 και θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Προεδρία. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι θα είχαν να πού οι δύο εισηγητέ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε το σημείο 11 και την πρώτη και να τελειώσουμε με αυτό το σημείο να ακούσω και να ακούσουμε μερικά συμπεράσματα. Να δώσω το λόγο στην πρώτη κυρία και μετά να δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν και να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα. Αυτά είναι καλύτερα να τα κάνουμε κάπως ε, χαλαρά. Όχι να προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε τη συζήτηση ε, περί Σέγγεν μέχρι τις 11.30. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή για τα διάφορα σημεία που εφήγησα μεταξύ των άλλων για να ενισχυθούν τα όσα κάνουμε. Παρόλα αυτά με απασχολεί η κατάσταση που αφορά τους ανήλικους. Δεν άκουσα να γίνεται αναφορά σε αυτό το θέμα, άκουσα την απάντηση της Επιτροπής και περίμενα μερικές πληροφορίες, αλλά δεν άκουσα τίποτα καινούριο οι ανήλικοι που έφτασαν στην Ευρώπη είναι όλο και περισσότεροι και θα μπορούσε αυτό να αιτιολογεί στην υιοθέτηση ενός ε, σχεδίου δράσης για τους ανηλίκους. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες συστάσεις προς τις χώρες μέλη σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν ε, και να ενσωματωθούν στα συστήματα. Η Έχω την εντύπωση ότι τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι αποδυναμωμένα. Χρειάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα ήθελα επίση να έχω περισσότερε πληροφορίε για το μηχανισμό επανεγκατάσταση όταν υπάρχουν ανήλικοι, όχι μόνο μη ασυνόδευτοι ανήλικοι. Το τελευταίο σημείο θα ήθελα να γνωρίζω αν στα πλαίσια αυτού του προγράμματο επαναπατρισμού από τη στιγμή που θα επιστρέψουν οι άνθρωποι στη χώρα του ελέγχεται το κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις γίνεται παρακρισμός και ε, ε, ε, πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης. Ευχαριστώ. Uh, Ο κ. Μισελ τώρα για να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών. Ευχαριστώ πρόεδρε για την πρώτη ερώτηση. Αλλαγή του Σέγγεν. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τι κάνουν τα κράτη αν έχει εκδοθεί η απόφαση η απόφαση απόφαση ε, επιστροφής χωρίς ή με βιομητρικά δεδομένα. Μπορούμε να υποβάλουμε περαιτέρω τροποποίηση στο πρωτόκολλο, αργότερο ωστόσο. Στο επόμενο σημείο για την ε, στελέχωση της υπηρεσία συζητούμε το ενδεχόμενο αύξηση του προσωπικού και της φρόνταξης και της ΕΑΖΟ και της Europol, αλλά μιλούμε για χαμηλά νούμερα. 60 τη Frontex, 40 για την ΕΑΖΟ, πρόκειται για αρχικά στοιχεία. Θα συζητούμε με, τη Γενική, με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και τους ανθρώπινους πόρους μας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η Frontex και η ΕΑΖΟ είναι εργαλεία για να διαμορφώσουν μέτρα με τα κράτη-μέλη. Η Frontex πρέπει να κάνει πρόσκληση εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη μέσω ενός συστήματος επιλογής εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη. Το ίδιο κάνει και η Άζο Στο hotspot, στο hotspot λοιπόν θα υπάρχουν υπάλληλοι προσωπικό του ΕΑΖΟ τη Frontex και αποσπασμένα στελέχη από τα κράτη-μέλη. Uh, Όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε από δικές μας δυνάμεις, ε, παίρνουμε στελέχη από τα κράτη-μέλη. Για τις επιστροφές, Προφανώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής επιστροφής. Προβλέπεται από την οδηγία. Δεν έχουμε λοιπόν μόνο την οικειοθελή αλλά και την υποχρεωτική επιστροφή. Η εθελούσια και μόνο δεν αρκεί γιατί σε μια περίπτωση το ποσοστό επιστροφή, το ποσοστό επιστροφών είναι πολύ χαμηλότερο. Βεβαίω οι επιστροφέ γίνονται σεβόμενοι τι διεθνεί αρχέ ε, και υποχρεώσει. Η Frontex ε, ε, έχει κονδύλια με καθαρά ε, αναλογικό τρόπο για το hot spot και πώς λειτουργεί. Καταχώρηση, καταγραφή των μεταναστών, δακτυλοσκόπηση, screening από τη Frontex, αν το άτομο ανήκει σε εθνικότητα με εξαιρετικά χαμηλό βαθμό αναγνώρισης και δεν ζητά άσυλο, μπαίνει στη διαδικασία επιστροφής. Αν είναι άτομο που έχει σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, μπορεί να μπει είτε στη διαδικασία ασύλου κανονικά ή στην διαδικασία με την κατάσταση, με ή άλλες εθνικότητες που αναφέρθηκαν. Έτσι θα λειτουργεί το hotspot. Για το... Για αυτούς που λένε ψέματα ως προς την εθνικότητα ή την ταυτότητά τους. Ο κόσμος, οι εργαζόμενοι εκεί έχουν εκπαιδευτεί για να διαπιστώσουν την εθνικότητα. Έχουμε διερμηνείς που μπορούν να δουν κατά πόσον ένα άτομο μιλά αραβικά με συριακή ή με μαροκάνικη προφορά. Υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχει Υπάρχει σύρος. Δηλαδή έχουμε και σύρους διερμηνείς. Στους ομαλούς είναι λίγο, στους είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί μιλούν γλώσσα κοντινή με τα τυγκρίνη που είναι της γειτονικής αιθιοπικής περιοχής. Υπάρχει όμως μια εκπαίδευση για να καταλάβει αν κάποιος είναι ερυθρέος ή όχι. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να καλύψουμε στα hot stop και να δούμε κατά πόσον οι ίδιες υπηρεσίες ασύλου στα κράτη-μέλη έχουν άτομα που μπορούν να ελέγξουν την προέλευση των ετούντων. Έχουμε plan B? Όχι. Πρέπει να εγκριθεί πρώτα πρώτα το πρόγραμμα και ζητώ από εσάς να, να βοηθήσει την εγκρισή του. Αυτό δεν είναι plan B, είναι plan A. Τώρα το θέμα του, της παρουσίας στρατού στα σύνορα. Ο κώδικας σύνορων Σέγγεν δεν αναφέρεται στο ποιο φυλάσσει τα σύνορα. Κάθε κράτος έχει διαφορετική, ε, διαφορετικά συστήματα. Ε, σε κάποια κράτη υπάρχουν σύνοριοφύλακες που ανήκουν στο στρατό ή είναι πολιτική υπηρεσία. Αυτό είναι θέμα όμως του κράτους μέλου Αυτό που χρειάζονται είναι σωστή κατάρτιση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τον σωστό τρόπο. Μπορεί να ανήκουν στο, να είναι στρατιωτικό σώμα, με θωριακή φρουή που ανήκουν στο στρατό δηλαδή. Ήδη, η συζήτηση, ήδη έγινε η συζήτηση της ασφαλές χώρες προέλευσης, αλλά ξαντεύχει το ερώτημα γιατί ευρωπαϊκή και όχι εθνικέ λίστε. Γιατί, μόνο γιατί να μην έχουμε μόνο ευρωπαϊκή λίστα και να έχουμε και εθνικέ. Σιγά σιγά εμείς υποβάλαμε μια ευρωπαϊκή λίστα, έναν ευρωπαϊκό κατάλογο στο, πρώτο, στο δεύτερο πακέτο ασύλου και απορρίφθηκε από το Συμβούλιο. Αν καταφέρουμε σταδιακά να επεκτείνουμε τον ευρωπαϊκό κατάλογο, ελπίζω κάποια στιγμή να μην χρειάζεται ο εθνικός κατάλογος, αλλά ας γίνει βήμα-βήμα. Δεν θα πετύχετε τώρα στο Συμβούλιο συμφωνία. Ιδίω διότι επικεντρωνόμαστε σε 7 χώρες και Υπάρχουν και άλλες χώρες που μπορεί να είναι σε εθνικό κατάλογο. Σταδιακά λοιπόν, ας προχωρήσουμε με τις πιο προφανείς περιπτώσεις τώρα και αν προχωρήσουμε αργότερα θα μπορούμε ίσως σε κάποια μεταγενέστερη φάση να εγκαταλείψουμε αυτούς τους εθνικούς καταλόγους. Το ποσοστό επιστροφών στην Ευρώπη είναι συνολικά για όλες τις εθνικότητες 40% όχι μόνο για τους ιεροκοινούς, για τους ανήλικους στο σύστημα με την κατάσταση υπάρχει σαφής αναφορά λήψη υπόψη της τροτότητας του ατόμου να ληφθούν υπόψη ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που μετεγκαθίστανται θα αντιμετωπιστούν με ειδική προσοχή, θα ληφθούν υπόψη περισσότερο οι προτιμήσει του κλπ. Αυτά και ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Τώρα αν κάποιος ε, πιστεύει ότι θέλει και άλλες λεπτομέρειες ε, στις ε, ερωτήσεις, προφανώς η Κομισιόν θα είναι στη διάθεσή του. Συνάδελφοι, όπως είπαμε, τα θέματα του Σέγγεν θα τα συζητήσουμε τον Οκτώβρη και έτσι θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι και κλεισμένων των κυρών. Να είναι σαφές ε, ότι τα μέλη άλλων επιτροπών, οι σύμβουλοι, οι βοηθοί θα μπορούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι σαφές ποιοι πρέπει να παρίστανται. Εκπρόσωποι του ΕΛΚ, Γενικός Γραμματέας, το προσωπικό της ΛΥΜΠΕ, εκπρόσωποι της νομικής υπηρεσίας του, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτοί είναι όλοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε 11.30 λοιπόν σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Μικρό διάλειμμα.